Sorry about that. I think this is a, an issue that's of great interest to those of... Καλημέρα σας. Νομίζω ότι το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις χώρες αυτές που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο πληθυσμό φωκών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η σχέση ανάμεσα στις φώκες και τα αλλιευτικά αποθέματα. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει τόσο επαγγελματίε του κλάδου όσο και επιστήμονες. Επίσης λέγεται ότι υπάρχει μία πολιτική διάσταση στο ζήτημα αυτό, τουλάχιστον για τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Αλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από, την, από το Τμήμα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διοργανώσει αυτό το εργαστήριο το οποίο θα ασχοληθεί ειδικά με το ζήτημα αυτό. Με ιδιαίτερη χαρά έχουμε σήμερα μαζί μας ένα πάνελ από αξιόλογους εμπειρογνώμονες οι οποίοι προετοίμασαν τέσσερις έρευνες για το ζήτημα αυτό. Οι έρευνες σας έχουν ήδη δοθεί, μπορείτε να δείτε κάποια αντίτυπα των μελετών που δημοσίευσαν οι προσκεκλημένοι μας. Τα τέσσερα άτομα λοιπόν, τα οποία είναι μαζί μας, θα ήθελα να τα καλωσορίσω και είναι ο κύριος Στέρο Χάρκνεν, ο οποίος θα ήταν ο πρώτος ομιλητής από το Σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Με ειδοποίησε ο κύριος Χάρκονεν ότι ε, έχει καθυστερήσει λόγω της ε, κίνησης. Έχουμε επίσης μαζί μας τον Φιλ Χάμον, το οποίος ήταν και ο πρώτος ομιλητής μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Μισελ Κρόνιν από το Πανεπιστήμιο του Κόρκ και τον κύριο Βέστεμπεργκ στο τέλος, ο οποίος εκπροσωπεί το Συνδικό Συμβούλιο Αλίας. Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Χάμον, θα ήθελα να σας πω ότι κάθε μιλητής έχει στη διάθεσή του 20 λεπτά και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και τον χρόνο στη συνέχεια μετά από κάθε παρουσίαση να κάνουμε συζήτηση, να υποβάλουμε ερωτήσεις. Επίσης θα ήθελα να σας πω για τα με τους βουλευτές από την Ιταλία που ενδεχομένω να είναι στην αίθουσα ότι τα Ιταλικά μεταδίδονται, η Ιταλική διερμηνία βρίσκεται πλέον στο κανάλι 4 γιατί η οθόνη που έχω από πίσω μου καλύπτει την ε, Ιταλική καμπίνα. Πρέπει λοιπόν να συνδεθείτε με την ε, καμπίνα επαριθμών 4 αν θέλετε να ακούσετε την Ιταλική διερμηνία. Δίνω ευθύ αμέσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Φίλιπ Χάμοντ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ βέβαια του ε, Συμβουλίου Θαλασσίων Θηλαστικών και του κυρίου Ιαν Μπόιντ από το Πανεπιστήμιο του Σαντ Άντριους θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση όπως έχει στην Σκοτία, ποια είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις φώκες και τα ελευτικά αποθέματα. Ήδη από τη δεκαετία του 1970 στα νερά της Σκοτίας παρατηρείται μια σημαντική μείωση των ελευτικών αποθεμάτων, ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι από τη δεκαετία του 1960 έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά ο πληθυσμός των φωκών. Βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι η βιομάζα των αλλιευτικών αποθεμάτων και πώς αυτή είχε εξελιχθεί από την δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα και πώς η μείωση αυτή συνδέεται με την αύξηση της, του πληθυσμού των φωκών. Βλέπετε για παράδειγμα πως η αρνητική μείωση στον γάδο συνδυάζεται με την θετική αύξηση στον πληθυσμό των φωκών. Είναι εύκολο πολύ να συνδυάσει κανείς αυτά τα δύο δεδομένα και να θεωρήσει ότι υπάρχει μια συσχέτιση. Στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Απλώ αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση του Ηνωμένου Βασίλειου και στη Σκωτία. Από την άλλη βλέπουμε ότι ο πληθυσμό των φωκών έχει παρουσιάσει αυξομοιώσεις. Είχαμε δύο σημαντικέ επιζωοτίε το 1988 και το 2002 που οδήγησαν σε μια προσωρινή μείωση του πληθυσμού των φωκών η οποία ακολουθήθηκε στη συνέχεια από μια σχετική αύξηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δύο σημαντικά νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με τι φώκες και την προστασία του. Η πρώτη είναι η οδηγία για τα ενδιατήματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σα εξηγήσω περισσότερο την οδηγία αυτή. Οι φώκε καλύπτονται από το παράρτημα επαναληφθμών 2, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργούν ειδικού χώρου προστασία για τι φώκε. Έχουμε όμω και ένα νέο νομοθέτημα στην Σκοτία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο προβλέπεται και μια προστασία για τις φώκες. Βάσει λοιπόν αυτών θα μιλήσω σήμερα το πρωί και θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες όσον αφορά τα αληφτικά αποθέματα, τα αποθέματα ηχθείων στην ε, Σκοτία, τον πληθυσμό των φωκών. Θα μιλήσουμε επίσης για την διατροφή των φωκών και ποια είναι η ε, επίπτωση που έχουν οι φώκες στα αληφτικά αποθέματα και θα, θα προσπαθήσουμε να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί και αυτό το ευρύτερο πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σύντομα τι είδου ε, ψάρια έχουμε στην ε, Σκοτία. Έχουμε καταρχάς αλία με τράτες βυθού. Χρησιμοποιεί τη μέθοδος αυτή κυρίως για τον γάδο, τον εγκλεφίνο, το νταούκι του Ατλαντικού, το μαυροπολάκιο. Έχουμε επίσης το βάτρα χόψαρο, την Μεσκαλτρίτσα, την οποία αλλιεύουμε. Επίση, ε, προσπαθούμε να αλλιεύσουμε κάποια είδη όπω το αμόχελο, το σίκο της Νορβηγία, την ρέγα και το σκουμπρί, κυρίως μέσω τη Αλλία μετράτας και χρησιμοποιούμε επίτα και τα σειρώμενα δίχτυα βυθού, κυρίως για καραβίδες και για το πλατύψαρο. Σαφώ χρησιμοποιούμε όμως και καλάμια καθώς επίσης και στάσιμα δίχτυα κυρίω για την αλίευση σολομού. Βλέπετε εδώ πέρα την αξία των αλλιευμάτων αυτό σε εκατομμύρια ε, λιρών. Βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσό έχουμε στις καραβίδες. Στη συνέχεια έχουμε το βατραχόψαρο, 28 εκατομμύρια λίρες. Δεν τρώνε βατραχόψαρο όμως οι φώκες. Και έχουμε και 58 εκατομμύρια λίρες που αντιστοιχούν κυρίως στην αλίευση γάδου εγκλεφίνου. Ήδη με τα οποία διατρέφονται όμως και οι φώκες. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μικρή επικάλυψη ανάμεσα στην αξία των αλλιευμάτων και τα αλλιεύματα εκείνα με τα οποία διατρέφονται κυρίω οι φώκε. Α αναφερθούμε τώρα στο ζήτημα κυρίω στην σχέση που υπάρχει μεταξύ Σολομού και φωκών στη Σκωτία. Και βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι η επίδραση που, μπορεί που μπορούν να έχουν κυρίω οι γκρίζε φώκε. Στην δεκαετία του 1990 τα περισσότερα αποθέματα Σολομού καθώς επίσης και ο πληθυσμός των φωκών παρουσίασε μείωση. Σε ορισμένε περιπτώσει θεωρήθηκαν οι φώκε υπεύθυνε για τη μείωση του σολομού και προχωρήσαμε σε κάποιου μεθόδου θανάτωσή του. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα διοδότησης που προβλέπεται στον νέο νόμο της Σκωτίας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Θα αρχίσει να ισχύει από το 2011 βέβαια και Το σύστημα προστασίας των φωκών που προβλέπεται στο νομοθέτημα αυτό ουσιαστικά βασίζεται σε ένα σχέδιο διαχείρισης που έχουμε από το 2005 και το οποίο ισχύει για την Ανατολική Σκοτία. Στόχος εδώ πέρα είναι να εξισορροπήσουμε τις ανησυχίες για την προστασία των ε, ειδών με, την, ε, με άλλες πολιτικές που μπορούν να έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την αλληλεία ή τον τουρισμό. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε κάποιες μεθόδους προστασίας, για παράδειγμα χρήση δικτυών γύρω από τις περιοχές αλίευσης ή ακόμα και κάποια ηχοακουστικά συστήματα αποθάρρυνσης των φωκών, αποτροπής των φωκών ή αν δεν λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά τότε προβλέπεται θανάτωση των φωκών με του φεκισμό αλλά και εδώ πέρα πάλι προβλέπονται συγκεκριμένα όρια. Δεν θα ήθελα να φερθώ περισσότερο τώρα στο ζήτημα του Σολομού και των φωκών. Το... Υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στα δύο αυτά ήδη. Η επίπτωση όμως των φωκών στον στα αποθέματα Σολομού είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Βλέπετε εδώ πέρα μία απλή αναπαράσταση των όσων πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε για τα λευτικά αποθέματα στην Σκοτία εδώ βασιζόμαστε κυρίως στην ε, βιομάζα που έχουμε για τα ίδια αυτά και κυρίως για την δυνατότητα, αναφερόμαστε κυρίως στη δυνατότητα παραγωγής των ειδών αυτών. Βλέπετε ότι για τα περισσότερα είδη είτε δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει γιατί δεν έχουμε αρκετά δεδομένα ή από ό,τι φαίνονται βρίσκονται σε καλή κατάσταση όσον αφορά τη δυνατότητα παραγωγής τους. Έχουμε πρόβλημα κυρίως με τον γάδο και αυτό ισχύει για τη Βόρεια Θάλασσα και τη Δυτική Σκοτία. Εδώ πέρα θεωρείται ότι υπάρχει χαμηλό επίπεδο αναπαραγωγή, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί. Η κατάσταση λοιπόν με τον γάδο δεν είναι καλή, γιατί τα υπόλοιπα είδη ή δεν γνωρίζουμε ή θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι καλή, αποδεκτή. Αν δούμε τώρα τα πράγματα στο ευρύτερο πλαίσιο του και δούμε πώ μπορούν να εξελιχθούν μακροπρόθεσμα, Εδώ ασχολούμεθα με τα επίπεδα που είχαμε στο παρελθόν και μπορούμε να βασιστούμε για ορισμένα ήδη ακόμα και στα δεδομένα που είχαμε από τη δεκαετία του 50 και του 60. Και σε όλε αυτέ τι μετρήσει που κάνουμε και σε όλε αυτέ τι συγκρίσει που γίνονται, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η βιομάζα αναπαραγωγή, δηλαδή το ποσοστό εκείνων των ειδών που είναι σε θέση να αναπαραχθούν και έχουμε έπειτα στη συνέχεια και τις εκφορτώσεις καθώς επίσης και τελευταία αποθέματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδίω όσον αφορά το σχετισμό τη βιομάζα με τελευταία αποθέματα, η βιομάζα παρουσιάζει αρκετά σημαντική μείωση. Επομένω, για πάρα πολλά είδη η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Α περάσουμε τώρα στι φώκε. Έχουμε δύο ειδών φώκε τη Σκοτία, στα νερά τη Σκοτία. Ο μεγαλύτερο πληθυσμό είναι τη γκρίζα φώκε που βλέπετε στα αριστερά σα. Ένα 40% του παγκόσμιου πληθυσμού γκρίζα φώκια ζει στη Σκοτία τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπε φώκε βρίσκονται στον Ατλαντικό, στον Καναδά κυρίω. Και έχουμε στη συνέχεια την Harbor Seal, την κοινή φώκια, που παρατηρείται και στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό. Στη Σκοτία έχουμε 25% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κοινή φώκια, Harbor Seal. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Σκοτία είναι μια σημαντική χώρα για αυτά τα δύο είδη φώκια. Κάποιε πληροφορίε για τα ίδια αυτά. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών κάνει επιτηρήσεις έρευνες από αέρος κάθε χρόνο και βλέπετε εδώ πέρα με διαφορετικά χρώματα την γκρίζα φώκια καθώς επίσης και την κοινή φώκια. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η κατανομή, η γεωγραφική κατανομή των δύο αυτών ειδών. Παρατηρούνται σε διάφορα σημεία της Σκοτίας. Υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, για παράδειγμα περισσότερες harbor φώκες στην περιοχή που βλέπετε εδώ πέρα στα δεξιά, στα δυτικά επίσης της Σκοτίας, στις δικές ακτές υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός κοινή φώκιας. Υπάρχει λοιπόν ένα διαχωρισμό, αν θέλετε, στην κατανομή. Υπάρχει όμω και μια αρκετά μεγάλη επικάλυψη, γεωγραφικέ ζώνες, δηλαδή, στις οποίε παρατηρούνται και τα δύο είδη. Επίση υπάρχουν. Ε, το, η γκρίζα φώκια περνάει περισσότερο καιρό στην ακτή, ακριβώ επειδή εκεί πέρα σε θέση να προσέχουν τα μικρά τους τους νεογνούς. Βλέπετε επίσης εδώ πέρα και την κατανομή της φώκιας στην θάλασσα. Όπως βλέπετε στην φωτογραφία αριστερά χρησιμοποιούμε κάποιους μικρούς πομπούς στο κεφάλι της φώκιας προκειμένου να καταφέρουμε να εντοπίσουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι φώκες 500 περίπου είναι οι φώκες οι οποίες έχουν... Όχι. Ε, έχουν το πομπό αυτό και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να δούμε πού ακριβώς βρίσκονται, σε ποια νερά ακριβώς ζουν. Οι ε, γκρίζες φώκες περνάνε περισσότερο χρόνο στην θάλασσα και βλέπετε κυρίως ποιες είναι οι περιοχές εκείνες στις οποίες στηρεύουν οι φώκες αυτές. Στα δεξιά βλέπετε την κατάσταση για την κοινή φώκια, Harbor Seal, εδώ πέρα η θήρευση είναι πολύ πιο ε, εντοπισμένη, πολύ πιο κοντά στις ε, ακτές. Οι φώκες αυτές ζουν πολύ πιο κοντά στις ακτές σε σχέση με τις ε, γκρίζες φώκες. Και γενικά μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι οι φώκες κυνηγούν κυρίως κοντά στις ακτές και κυρίως στα νερά. Όσον αφορά τώρα το μέγεθος του πληθυσμού, Κάθε φθινόπωρο κάνουμε έρευνες από αέρος, βγάζουμε φωτογραφίες σαν αυτή που βλέπετε στη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ πέρα μία φωτογραφία που δείχνει φώκες και νεογνούς σε έναν τόπο αναπαραγωγής. Και χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες αυτές για να καταφέρουμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό των φωκών που χρειάζεται για την ε, Αναπαγωγή την οποία βλέπουμε στη φωτογραφία. Βλέπετε εδώ πέρα τον συνολικό πληθυσμό, καθώς επίσης και τα στοιχεία που έχουμε από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα. Με διαφορετικά χρώματα βλέπετε τις διαφορετικές περιοχές της Σκοτίας, στις οποίες παρατηρούνται οι φώκες αυτές Orkney Hebrides. Στο Hebrides, για παράδειγμα, στην, με την μπλε γραμμή, βλέπουμε ότι ε, τα ποσοστά αναπαραγωγής στις φώκες έχουν μείνει σταθερά ή παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση, λιγότερο από 1% ετησίως. Επομένως, η γκρίζα φώκη, η οποία παρουσίαζε ε, αύξηση στον πληθυσμό της τελευταία χρόνια, παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια σταθερότητα, μια στασιμότητα. Όσον αφορά τώρα την Harbour Seal, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιες εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό φωκών που βρίσκονται στην ξηρά. Βλέπετε κάποιες εικόνες με θερμική επικόνωση. Βλέπετε εδώ πέρα τις φώκες με το λευκό χρώμα. Το σκούρο χρώμα είναι η θάλασσα. Κάνουμε λοιπόν έρευνες με ελικόπτερα το καλοκαίρι και χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες αυτές, τις έρευνες αυτές για να κάνουμε μια μέτρηση του πληθυσμού. Τη δεκαετία του 1990 το μέγεθος του πληθυσμού για διάφορες περιοχές της Σκωτίας με ένα σύνολο 29.000 ε, περίπου ε, φώκες. Σε άλλες περιοχές βλέπετε ότι στις αρχές του 2000 ή στη συνέχεια στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπάρχει μια σημαντική μείωση του πληθυσμού, ιδίως στο Όρκνη. Ο συνολικός πληθυσμός της Φώκης αυτή τη στιγμή στη Σκοτία που έχουν μετρηθεί στην ξηρά είναι γύρω στις, γύρω στις 20.000. Ο συνολικός πληθυσμός υπολογίζεται από τον χρόνο που περνάνε στην ξηρά και στη θάλασσα και μπορούμε να πούμε ότι και για τα δύο είδη φτάνουμε σε ενα αριθμο αριθμό 40-46.000. Συνοπτικά έχουμε 100.000 περίπου γκρίζες φώκες στην Σκοτία, σταθερός πληθυσμό μετά από πάρα πολλές δεκαετίες αύξηση και έχουμε περίπου 40.000 φώκες Harbor, κοινέ φώκες, που παρουσιάζουν έντονη μείωση στα βόρεια και στην ανατολικά και έχουν σταθερή ανάπτυξη στα δυτικά της Σκοτίας. Με τι διατρέφονται τώρα οι φώκες. Στη Σκωτία υπάρχουν δύο έρευνες για την ε, αξιολόγηση της διατροφής στις ε, φώκες. Το 1985 και το 2002 γίνανε δύο σημαντικές έρευνες. Βλέπετε τις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες ε, εντοπίστηκαν οι έρευνες αυτές. Όσον αφορά την ε, κοινή φώκη, για αυτήν δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και οι περισσότερες δεν είναι επικαιροποιημένες. Για την κοινή φώκη δεν γνωρίζουμε όσα γνωρίζουμε για την γκρίζα φώκια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει τώρα μια νέα έρευνα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Σκοτίας προκειμένου να καταφέρουμε να ερευνήσουμε περισσότερο την διατροφή την οποία την τάση διατροφή στην οποία ακολουθεί η γκρίζα φώκια. Πρέπει όμως να δούμε με τι διατρέφονται και τα δύο είδη για να δούμε αν ε, υπάρχουν κάποια ε, είδη αλλιευτικά τα οποία, με τα οποία διατρέφονται και οι δύο κατηγορίες. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες ε, εκτιμήσεις με ένα πολύ απλό τρόπο. Πηγαίνουμε ουσιαστικά στις ακτές μαζεύουμε τα απομεινάρια που έχουν απομείνει στην ακτή, από αυτά τα οποία έχουν φάει δηλαδή οι φώκες και προσπαθούμε από αυτά που έχουν απομείνει να δούμε τελικά με τι διατρέφονται οι φώκες. Μπορούμε να μετρήσουμε τα απομεινάρια αυτά και μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και τα δύο είδη φώκες. Σαφώς πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της ε, έρευνας, αλλά πιστεύω ότι για τις ε, γκρίζες φώκες και για την κοινή φώκες στη Σκωτία η μέθοδος αυτή έχει δώσει θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά δηλαδή την αξιολόγηση αποτίμηση των μεθόδων διατροφής. Βλέπετε εδώ πέρα τις έρευνες για το 1985 στα αριστερά και το 2002 στα δεξιά για τη δυτική ακτή του Όρκνη και την ανατολική ακτή της Σκωτίας. Με κίτρινο βλέπετε τα αμόχελα με μπλε τα γαδοειδή, όπου έχουμε τον γάδο, τον μελού και το προσφυγάκι. Έχουμε το πλατήψαρο στη συνέχεια. Με το πράσινο έχουμε τα πελογικά είδη, όπως ο μερλούκιος και το σκουμπρί. Βλέπετε ότι περισσότερες φώκες τρέφονται με ή γαδοειδή και έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές ανάμεσα στο 1985 και το 2002. Στη δική ακτή και στο Όρκνη η κατανάλωση αμόχελων έχει μειωθεί, αλλά στην ανατολική ακτή μεταξύ 1985 και το 2002 η κατανάλωση αμοχέλων έχει αυξηθεί. Για τα αγωδοειδή η κατάσταση έχει παραμείνει η ίδια, αλλά παρουσιάζει μείωση έχει αυξηθεί μάλλον στο Όρκνη και έχει μειωθεί στην Ανατολική Ακτή. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιφερειακές γεωγραφικές διακυμάνσεις όσον αφορά την κατανάλωση αμοχέλων γαδοειδών, που είναι και τα δύο βασικά είδη διατροφής της ε, φώκιας. Θα μπορούσαμε τώρα να ερμηνεύσουμε με ποσοστά, με αριθμητικά στοιχεία τα δεδομένα αυτά για, την, ε, για τη χωματίδα, το αμόχελο, τον γάδο, τον εγκελφίνο. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ποια είναι τα ακριβή ποσοστά που έχουμε για το 85 και το 2002. Για παράδειγμα, για τον γάδο Έχουμε 4.000 περίπου τόνους που έχουν καταναλωθεί το 1985 από γκρίζες φώκες, ενώ το 2002 ο αριθμός αυτός έχει γίνει 8.300 τόνοι. Βλέπετε ότι η συνολική κατανάλωση το 1985 38.000, το 2002 116.000. Η σημαντική αυτή αύξηση εξηγείται από το ότι τριπλασιάστηκε ο ρυθμός των φωκών μεταξύ 85 και 2002. Το σημαντικό είναι να δούμε εδώ πέρα το ποσοστό των τόνων αυτών όσον αφορά τα εμπορικά λιευτικά αποθέματα και όσον αφορά την συνολική βιομάζα των αποθεμάτων. Μπορείτε να δείτε για όλα αυτά τα ίδια ότι για το 1985 το ποσοστό το οποίο κατανάλωναν οι φώκες ήταν ε, χαμηλό, ενώ το 2002 έχουμε μια σημαντική αύξηση στα ποσοστά αυτά. Για τα περισσότερα είδη μπορούμε να πούμε το ποσοστό παραμένει χαμηλό, παρόλα αυτά για κάποια είδη όπως ο γάδος έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Επομένως, η θνησιμότητα για ορισμένα αλλιευτικά είδη που προκαλείται από τις φώκες αρχίζει και γίνεται πλέον στατιστικά σημαντική. Επίσης, βλέπετε εδώ πέρα ότι η κατανάλωση αναφώκη είναι 5 κιλούς, 5 κιλά 5 κιλά ημερησίως. Βλέπετε εδώ πέρα την κατανάλωση πιο συγκεκριμένα για την γκρίζα φώκια. Πάλι στοιχεία 1985 και 2002. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το ποσοστό που καταναλώνεται από την γκρίζα φώκια είναι σημαντικότερο σε σχέση με την κοινή φώκια. Και βλέπετε το 300% το φοβερά μεγάλο αυτό ποσοστό για το 2002 που αντιστοιχεί στο ποσοστό αλληλευτικών αποθεμάτων που έχει ε, καταναλωθεί από φώκες. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιό τους. Δεν έχουμε πάρα πολλά αντικειμενικά στοιχεία από τις δυτικές ακτές της Σκοτίας. Σίγουρα οι φώκες αποκλείεται να καταναλώνουν τόσο μεγάλα ποσά και το ποσοστό αυτό σίγουρα δεν είναι αντικειμενικό, αλλά σίγουρα συμβάλλουν στην ε, κατανάλωση. Αυτέ είναι οι πληροφορίε που έχουμε μέχρι στιγμή. Από ό,τι φαίνεται, οι φώκε τρέφονται κυρίω με ε, προσφυγάκι, ρέγγε, αμόχελα. Δεν είναι επικυρωποιημένα όμω τα στοιχεία αυτά. Ανταποκρίνονται περισσότερο στη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Συνοψίζοντα, μπορούμε να καταλήξουμε στο εξή συμπέρασμα, ότι οι γκρίζε φώκε καταναλώνουν 100.000 τόνου ε, τον χρόνο, κυρίω αμόχελα και γαδοειδή, ενώ η κοινή φώκια, η Harbour Seal, καταναλώνει περίπου 80.000 τόνου τον χρόνο, κυρίω αμόχελα, γαδοειδή και ρέγγε. Νομίζω θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να δούμε και ποιοι είναι οι άλλοι κυνηγοί, ποια είναι τα άλλα αρπακτικά, αν θέλετε, που καταναλώνουν ε, ψάρια. Είπαμε ότι οι φώκε καταναλώνουν περίπου 270.000 τόνους ψάρια το χρόνο. Μπορούμε ανάλογου υπολογισμού να κάνουμε και για τα κοιτοειδή, δηλαδή τα δελφίνια, κυφάλαινες, που καταναλώνουν 300.000 τόνους, πάνω κάτω τα ίδια δηλαδή με τις φώκες. Στη συνέχεια έχουμε τα θαλασσοπούλια και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βασική κυνηγή ψαριών είναι τα άλλα, τα μεγαλύτερα ψάρια τα θαλασσοπούλια καταναλώνουν 600.000 τόνους ψαριών των ετησίως, ενώ τα υπόλοιπα ήδη τα ψάρια, καταναλώνουν 2 εκατομμύρια τόνους ετησίως ψαριών. Βλέπετε εδώ πέρα ποιε είναι οι επιπτώσεις δηλαδή από τους κυνηγού αυτούς, από τη θύρευση αυτή στα λευτικά αποθέματα. Αν δούμε λοιπόν τις φώκες στο ευρύτερο πλαίσιό τους, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντική κυνηγή τελικά ψαριών και ότι δεν συμβάλλουν τόσο πολύ στη μείωση των ελευτικών αποθεμάτων. Καταλήγουμε λοιπόν στα συμπεράσματα τα ακόλουθα. Σαφώ τα ελευτικά αποθέματα στη Σκωτία παρουσιάζουν μείωση κάτω από τα ιστορικά επίπεδα. Ο πληθυσμό τη ε, γκρίζα φώκες έχει σταθεροποιηθεί, ενώ τη κοινή της τη Σιλ έχει παρουσιάσει μείωση τελευταία δεκαετία. Επίση υπάρχει σημαντική επικάλυψη ανάμεσα στη θύρευση που γίνεται από τις φώκες και την αλία. Παρόλα αυτά, ε, τα ποσοστά ε, μείωσης των ελεκτικών αποθεμάτων που οφείλονται στη θύρευση από φώκια είναι πολύ μικρότερα από τα ποσοστά εκείνα που έχουν να κάνουν με, την, με τον ανθρώπινο παράγοντα, με την αλία πιο συγκεκριμένα και όπως εξηγήσαμε πριν από λίγο η επιρροή της φώκιας αν δούμε την συμμετοχή της στο ευρύτερο πλαίσιο είναι πολύ πιο χαμηλή από ό,τι θα περίμενε κανείς δηλαδή αν συγκρίνουμε τη φώκια με τους υπόλοιπους θηρευτές ψαριών. Και ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό ότι η επίπτωση δηλαδή από τις φώκες είναι πολύ μικρότερη όσον αφορά τα συνολικά ποσά αληφτικών αποθεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε, ιδιαίτερα επειδή εγώ προέρχομαι από την Σκοτία ίσως. Και πράγματι συνάδει και με τις, αυτά που είπατε συνάδουν και με τις πληροφορίες που είχα ακούσει και στο παρελθόν. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα. Ο κύριος Τέρο Χάρκενεν είναι εδώ. Ωραία λοιπόν. Ας του δώσουμε το λόγο από το Σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τον καλωσορίζουμε στη συνεδρίασή μας και θα, το θέμα του είναι φώκες και αλληλευτικά αποθέματα στον βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό. Κύριε Χάρκενεν, έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε. Thank you um, Ευχαριστώ πολύ θα κάνω μια παρουσίαση για τον πληθυσμό των φωκών, για την διατροφή τους, για τα παράσιτα των φωκών και για την επίδρασή τους στο περιβάλλον και στα αποθέματα. Θα αναφερθώ σε μια-δυο περιοχές και στη Βαλτική. Έχουμε πληροφορίες από την Ισλανδία, από τη θάλασσα του Μπάρεντς και από την ε, δυτική όπτη της Νορβηγίας. Αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την Ιρλανδική θάλασσα και για τη Σκοτία. Και αρχίζω με τα είδη των φωκών. Όπως είπε και ο Φιλ, υπάρχουν δύο είδη κυρίως στο βορειοανατολικό Ατλαντικό η γκρίζα φώκια και η κοινή φώκια, harbor seal. Αλλά υπάρχουν και οι ριγέ φώκε, ringed seals, στη Βαλτική αλλά και στην Αρκτική θάλασσα ζουν αυτές. Υπάρχουν μετά και οι harp seals, η λευκότριχη γρυλανδική φώκια, φώκια της ε, Γρυλανδίας, στη θάλασσα του Μπάρεντς και το 1987 ήρθαν στην ε, προσέγγισαν την δυτική ακτή της Νορβηγίας και ε, προξένησαν ζημιές στην Αλία. Βεβαίως, οι φώκες επηρεάζουν τα λευτικά αποθέματα, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των φωκών, από τη διατροφή τους, από την ποσότητα που τρώνε και από τα ίδια τα αλλιευτικά αποθέματα και τη μορφή που έχουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Θα δούμε βέβαια πώς επηρεάζονται αυτά τα αλλιευτικά αποθέματα από τις φώκες σε διάφορες χώρες. Αν δούμε την ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή τα ωκεάνια συστήματα, θα δείτε ότι εκεί η θνησιμότητα που οφείλεται στις φώκες είναι κάτω από 1% των αποθεμάτων αναπαραγωγής των ψαριών. Σε αυτά τα συστήματα λοιπόν, αν αφαιρέσουμε θεωρητικά τον πληθυσμό των φωκών, δεν θα άλλαζε και τίποτα ούτε η αλία θα βελτιωνόταν, τα αλλιεύματα δηλαδή. Αλλά σε ορισμένα από αυτά τα συστήματα, όπως παραδείγματος αν στη θάλασσα του Μπάρεντς, τα αποτελέσματα των φωκών είναι πιο έντονα. Γιατί υπάρχουν δύο εκατομμύρια harp seals εκεί. Ε, άρα σημαντικό ποσοστό του οικοσυστήματος είναι η φώκη αυτή της Γρυλανδίας, hard Seals. Ε, φτιάξαμε μοντέλα τα οποία μελετήσαμε και είδαμε ότι αν αλλάξουμε λιγάκι τη διατροφή όσον αφορά το γάδο ε, και εκεί δεν επηρεάζονται τα πράγματα πολύ δεν ε, παθαίνει τίποτα ο πληθυσμό φώκια, δηλαδή αν δεν υπάρχει αρκετός γάδος. Εδώ βλέπετε την κοινή φώκια στη Δανία, στη Γερμανία και αυτές οι, και αυτή η κοινή φώκια ε, ζει κοντά στην ε, ακτή συνήθως, αλλά βεβαίω, καμιά φορά κυνηγάει και πιο μακριά από την ακτή. Σε αυτά όμως τα παράκτια τα συστήματα, δεν μιλάμε πια για τα ωκεάνια, μιλάμε για τα παράκτια συστήματα, όχι στην ανοιχτή θάλασσα. Εδώ ίσως είναι πιο μεγάλη η επίδραση της φώκιας στα ενδυνάμει, στα τοπικά αποθέματα. Όμως η... για ορισμένα αποθέματα είναι πιο έντονη η επιρροή. Παραδείγματο χάρη στα εκβολέ ε, των ποταμών Σκοτία, τέτοιου είδου συστήματα. Βεβαίω, όπω ακούσατε, επηρεάζεται ο Σολομό στη Βαλτική θάλασσα. Είχαμε μείωση κατά 20% περίπου στα αποθέματα Σολομού λόγω της φώκιας εκεί, στη Βαλτική. Αλλά βεβαίως αυτά τα, αυτές οι επιδράσεις δεν είναι εύκολο να τις αποδείξουμε, να τις καταδείξουμε. Γιατί, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ α, πολλά άλλα αρπακτικά ψάρια σε αυτά τα συστήματα και αυτά τα άλλα ψάρια είναι πολύ περισσότερα σε αριθμό και καταναλώνουν, τρώνουν μεγαλύτερες ποσότητες από τη φώκες. Using tools and uh, other active... Τώρα, για τα αλλιευτικά εργαλεία. Υπάρχουν τα ενεργητικά και τα παθητικά αλλιευτικά ε, εργαλεία. Τα, τα ενεργητικά επηρεάζονται πάρα πολύ λίγο από τις φώκες. Βεβαίως υπήρξαν ε, καταγγελίες ε, γιατί μπερδεύονται οι φώκες πολλές φορές σε αυτά τα ενεργητικά αλλιευτικά εργαλεία. Και επηρεάζουν τα κύρια αλλιεύματα αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό για τα ενεργητικά αλλιευτικά εργαλεία και στην ανοιχτή θάλασσα λοιπόν δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αντίθετα στη παράκτη αλία και στη, στα στατικά αλλιευτικά εργαλεία, τα παθητικά αυτά τα bagnets, gillnets, αυτού του είδους τα δίχτυα, εκεί πραγματικά η φώκια επηρεάζει αρνητικά. Βεβαίως αυτά τα εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται ευρέω στο βόρειο Ατλαντικό, στο Ανατολικό Ατλαντικό. Χρησιμοποιούνται στη Βαλτική κυρίω και σε κάποιε παράκτιε περιοχέ, διότι δεν είναι ιδιαίτερα ε, κατάλληλα για αλεία σε περιοχές με έντονη παλήρια. Ωστόσο, πραγματικά οι φώκες ε, ε, επιτίθενται αν θέλετε σε αυτά τα στατικά εργαλεία για να πάρουν βέβαια το αλίευμα και στη Βαλτική θάλασσα έχουν πυροβοληθεί οι φώκες Α, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάσει θετικά την κατάσταση Επίσης οι φώκες έχουν παράσιτα τα οποία διαχέουν στο περιβάλλον. Τα σκουλίκια της φώκιας, seal worms, είναι το πιο ε, σημαντικό παράσιτο και στη θάλασσα του Μπάρεντς 95 με 96 τα 100 των αποθεμάτων κάποιων γαδοειδών και γάδου ε, έχουν μολυνθεί από αυτά τα σκουλίκια αλλά εκτός από τα σκουλίκια της φώκες υπάρχουν τα σκουλίκια της φάλαινας whale worms και η μόλυνση προέρχεται από τα δύο είδη αυτά σκουλικιών. Από εκεί και πέρα βεβαίω πειράζονται και μολύνονται και άλλα ε, αλλιευτικά άλλα είδη ψαριών. Εδώ προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μελέτη για το... και πήραμε δείγματα από διάφορες περιοχές που βλέπετε εδώ, από πολλούς ε, επιμέρους πληθυσμούς γάδου για να δούμε τα ποσοστά μόλυνσης από παράστα και βλέπετε σε αυτόν εδώ τον ε, πίνακα το A-Simplex είναι ο, το σκουλίκι της φάλαινας και το P-Decipiens είναι της φώκιας. Βλέπετε λοιπόν εδώ πώς επηρεάζονται τα πράγματα και προφανώς το whale worm, asimplex, είναι αυθονή σε όλες τις περιοχές εκτός από το φιόρ του Τρόνχαϊμ. Αντιθέτως, τα παράστα της φώκιας αυθονούν μόνο στην Ιρλανδική θάλασσα και στη Βόρεια θάλασσα στο Σκαγεράκι. Ε, σε γενικές γραμμές όμως τα τα δείγματα από την ανοιχτή θάλασσα δείχνουν μικρή μόλυνση ενώ τα παράκτια δείγματα δίνουν υψηλή ε, μόλυνση από το P. decipiens που είναι το λεγόμενο seal worm. Ένα συμπέρασμα λοιπόν που μπορούμε να εξάγουμε είναι ότι το σκουλίκι της Φώκιας δεν επηρεάζει πολύ τα αλλιεύματα της ανοιχτής θάλασσας. Αντιθέτως, για ψάρια τα οποία αλλιεύονται κοντά στην ακτή και κοντά στις ε, ε απικίες ε, φώκιας, εκεί που ζουν οι φώκιες κοντά στην ακτή, επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Βεβαίως, για να διαδοθούν τα παράστατα αυτά πρέπει να υπάρχουν και διάμεση ξενιστές κυρίως ασπόνδυλοι και πολλές, ε, πολλούς από αυτούς τους ξενιστές δεν τους βρίσκουμε στα, στις περιοχές των εκβολών ποταμών, των Δέλτα. Κάποια ήδη βεβαίως ε, κάποιοι ξενιστές ας πούμε τρώνε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες γόνου, λάρβας ε, του σκουλικιού αυτού και όταν φαγωθούν κατόπιν από το γάδο προφανώς προκανούν σημαντική μόλυνση. Αλλά σε γενικές γραμμές ε, το σκουλίκι της φώκιας δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Τώρα, η υδροκαλλιέργεια, η δατοκαλλιέργεια, ε, η οποία αυξάνεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, σχεδόν ένα εκατομμύριο ο, ψαριών ε, παρήχθη βλέπουμε στην Νορβηγία και στην, ε, δεν έχουμε στοιχεία για την Ισλανδία αλλά στις νήσες Φάροες στις Φαρόες νήσους υπάρχουν ε, καλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες και όλες αυτές οι υδατοκαλλιέργειες, αυτές οι φάρμες, οι ηχθειοκαλλιέργειες, ε, εκμεταλλεύσεις αυτές ε, αυτές τις επισκέπτονται οι φώκες και μπορούν να τις επηρεάσουν. Και στη Σκοτία βλέπουμε να επηρεάζονται. Μέχρι. Κυρίως στη Σκοτία με, που φτάνει μέχρι 5% η επιρροή. Αλλά σε όλες τις άλλες περιοχές τα ποσοστά είναι μικρά, είναι κάτω από 1%. Τι κάνουν ε, οι χθεοκαλλιεργητές πυροβολούν, πυροβολούν στη, τις φώκες εκεί. Βεβαίω απικίες φώκες δεν υπάρχουν στα, ε, στα φιόρδα αυτά που αναφέρουμε εδώ, Νορβηγία, Φαρόες και τα λοιπά, αλλά ε, γίνεται, πυροβολούνται οι φώκες και μάλιστα ε, συχνά και φαίνεται να θεωρείται ότι ε, τα αποτελέσματα είναι καλά. Το ίδιο γίνεται και στη Σκωτία. Πυροβολούνται οι φώκες, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τη Σκανδιναβία. Στις ε, λοιπόν αυτές δημιουργούν ζημιές οι φώκες, οι οποίες είναι μικρές όμως οι ζημιές αυτές. Πάντως η αντίδραση των ηχθειοκαλλιεργητών είναι να πυροβολούν τις φώκες για να μειώσουν το αποτέλεσμα. Στη σκοτία χρησιμοποιούνται και ε, ακουστικά αποτρεπτικά μέσα. Μερικοί λένε ότι τα αποτελέσματα είναι καλά, μερικοί λένε πως όχι. Δεν είναι σαφή η αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων. Για να κλείσω όμως την παρέμβασή μου, να εξάγω κάποια συμπεράσματα, να πω ότι η κατανάλωση των ε, φωκών ε, συνίσταται σε ένα ποσοστό κάτω από 1% των αλλιευμάτων. Ε, από τα αλλιευτικά αποθέματα ή από τα αποθέματα αναπαραγωγής. Με άλλα λόγια είναι άνευ σημασίας, μηδαμινή σημασία στα ωκεάνια συστήματα ή ζημιές από τη φώκια. Από εκεί και πέρα, γύρω στο 90% της αλίας ε, στο νοτιοανατολικό Ατλαντικό γίνονται με ενεργητικά ε, εργαλεία και εδώ πάλι η επίδραση της φώκιας είναι μηδαμινή. Πολύ μικρή. Βεβαίω ε, ζημιές υπάρχουν στα εργαλεία αυτά καθε αυτά. Είναι μικρή στα αποθέματα, η επίδραση τη φώκε, αλλά οι ζημιές στα εργαλεία μεγάλα. Από εκεί και πέρα, κυριω η αλία γίνεται με στατικά αλλιευτικά εργαλεία και εκεί η επίδραση μπορεί να θεωρηθεί μεγαλύτερη. Για τα στατικά εργαλεία λοιπόν, για τα ε, nets και τα bag nets που έλεγα προηγούμενα για αυτού του είδους τα δίκτυα. Ε, είναι, υπάρχουν ζημιές, ιδιαίτερα τα, για τα gill nets, ε, είναι πολύ δύσκολο να προστατευθούν και για τα μπάγκνετ, σας πούμε που χρησιμοποιούνται για την αλία χελιού και αυτά επηρεάζονται οι στατικές παγίδες για κάποια είδη ψαριών, για τα χέλια κυρίως και αυτά επηρεάζονται από τις φώκες αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Για την ανοιχτή θάλασσα τώρα ζημιές ε, και απώλειες πολύ μικρότερες από ό,τι για την παράκτη αλία και, γιατί, και όσον αφορά τα πατημόλυνση από τα παράσιτα. Πολλές φορές το σκουλίκι της φώκιας μπερδεύεται, γίνεται σύγχυση με το σκουλίκι της ε, φάλαινας. αλλά το, όπως σας είπα το σκουλίκι της φώκιας δεν ε, δημιουργεί τεράστιες απώλειες και τεράστια μόλυνση. εκείνο που μπορούμε να συμπεράσουμε εδώ βεβαίως, επειδή πυροβολούν πολύ τις φόκες, είναι να πούμε ότι ε, τελικά όντως ε, ο πυροβολισμός της φώκιας έχει αποτελέσματα τα πράγματα είναι διαφορετικά στις διάφορες γεωγραφικές περι περιοχές. Βέβαια σε περιοχές όχι απλώς μειώθηκε ο πληθυσμός της φώκες αλλά ε, εξαφανίστηκαν σχεδόν οι φώκες και εδώ παίζει ρόλο η ε, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στη διατήρηση των θαλασσίων θηλαστικών που πρέπει να προσεχθεί. Αντίστοιχα αναφέρεται Φέρονται αυτά και στις ε, συστάσεις της Επιτροπής του Ελσίνκη του 2006 ότι πρέπει να προστατευθούν για όλους αυτούς τους λόγους ίσως οι φώκες σε κάποια γεωγραφικές περιοχές. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ κυρία Χαρκόνεν. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Μισελ Κέρνεν που θα μας μιλήσει για την Ιρλανδία. Η κυρία Κρόνεν, συγγνώμη, σας δίνουμε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη τιμή είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω το θέμα αυτό της φώκες και των ελευτικών αποθεμάτων στα Ιρλανδικά. Είδατε, εργάζομαι στο Cork, στο University College. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους Gisop και Reed που με βοήθησαν να προετοιμάσω την ομιλία μου συνοπτικά γιατί θα σας παρουσιάσω, γιατί θα σας μιλήσω σήμερα. Τα κύρια στοιχεία της ομιλίας μου λοιπόν αφορούν πρώτα απ' όλα τις ε, φώκες, τον πληθυσμό φώκες στην ε, Ιρλανδία, τον αριθμό τους, την κατανομή τους και την διατροφή τους. Θα σας μιλήσω γενικότερα για την αλληλεία στην Ιρλανδία και την αλληλεπίδραση. Θα δούμε πώς επηρεάζεται γενικότερα η αλληλεία από την ύπαρξη της φώκιας και ποια είναι τα μέτρα ελέγχου που λαμβάνονται για την φώκια και για τα άλλα αρπακτικά ποια είναι τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις δεδομένων, κενά δεδομένων και θέματα διαχείρισης τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα κάνω και κάποιες συστάσεις στο τέλος. Λοιπόν, ποιες είναι οι φώκες που βρίσκομαι στα δικά μας τα ύδατα. Η γκρι φώκια και η Grey Seal και η Harbor Seal, η κοινή φόκια που είναι περισσότερο στον βόρειο ε, ε, Ατλαντικό. Τα ε, η λατινική τους ονομασία χάλι κόρους γκρίπους και Φόκα βιτουλίνα. Μιλώντας τώρα για τον διάφορα ίδια, είδη τα οποία έχουμε και για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο. Θα σας πω ότι οι κοινέ φώκες, στις, για τις κοινέ φώκες έγινε μια απογραφή σε βάση. Μια στιγμή, τη στιγμή την οποία έρχονται προς την ακτή όλες οι φώκες. Εδώ βλέπετε πώς έχουν εμφανιστεί στην ακτή της ε, Ιρλανδίας όλες οι φώκες. Έχουμε ε, χρησιμοποιήσει δηλαδή ε, με ελικόπτερο την τεχνική της φωτογράφησης για να μπορέσουμε να μετρήσουμε πόσες είναι. Είναι σημαντικό να δούμε ότι βεβαίως δεν μπορούμε να μετρήσουμε όλες τις φώκες. Έχουμε λοιπόν κάποιες ελίξεις. Έχουμε λοιπόν εκτιμήσεις ε, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό φωκών. Όσον αφορά τώρα τις γκρι φώκες. Η απογραφή έγινε κατά την διάρκεια της εποχής παραγωγής. Αναπαραγωγής τους μετρήσαμε όλα τα μωρά φώκες που βρέθηκαν στις ακτές. Παίρνοντας πάλι αεροφωτογραφίες και έχουμε ένα στατιστικό πρότυπο το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την μέτρηση και προσπαθούμε να μετρήσουμε την παραγωγή και, τον, ε, και να μετρήσουμε τα μωρά της φώκιας για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις εκ των υστέρων. Τώρα, η πρώτη σφαιρική απογραφή και μέτρηση έγινε στην Ιρλανδία αρκετά πρόσφατα το 2003 σε όλες τις ακτές. Σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις είχαμε λιγότερα από 3.000 ε, θηλαστικά φόκερ σε, όλη την, σε ελάχιστο αριθμό. Σε όλη την Ιρλανδία έχουμε περίπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, 4.000 Πάλι σας λέω ότι πρόκειται για εκτίμηση του ελάχιστου αριθμού αυτών των θηλαστικών, διότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε με ακρίβεια όλες. Περίπου δηλαδή έχουμε μετρήσει, φαντάζομαι, το 60 με 70% των θηλαστικών, τα οποία φτάνουν μέχρι τις ε, ε ακτές. Πρόκειται λοιπόν για... Ε, χοντρικά, αν θέλετε, αποτελέσματα, διότι δεν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιόπιστα για τον συνολικό αριθμό. Φαντάζομαι ότι στο σύνολο θα μπορούσαμε να πούμε ότι χοντρικά ότι έχουμε γύρω στις 7.000. Τώρα, το 2, για την κρή φώκια έγινε το 2005 μία απογραφή των ε, μικρών ε, θηλαστικών, των μωρών φώκες. Περίπου λοιπόν εκτιμήσαμε ότι γεννήθηκαν το 2005 1574 μωρά φώκες. Μέτρηση έγινε κυρίως στην Δυτική Ακτή. Άρα πιστεύουμε ότι στο σύνολο έχουμε περίπου ε, όλων των ηλικιών γκρι φώκες 5,5 με 7.000. Ποιες είναι οι τάσεις που διαγράφονται. Δεν έχει ε, γίνει καμία αξιολόγηση των τάσεων. Βασιστήκαμε μόνο στις εκτιμήσεις τις οποίες κάναμε το 2003 και το 2005. Δεν έχει γίνει από τότε μέχρι τώρα καμία ε, μελέτη εκτίμηση ε, μέχρι σήμερα για να δούμε αν αυξομειώνονται ε, τα θηλαστικά. Έχουμε βεβαίως ε, αποδείξεις ότι έχουν ε, αυξηθεί στην νοτιοδυτική Ιρλανδία οι κοινέ φώκες σε ποσοστό 13% το 1985 και 2006 ενώ τα μωρά φώκιας έχουν αυξηθεί στην ίδια περιοχή νοτιοδυτική κατά 50% από το 2003. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία ε, μελέτη σε εθνικό επίπεδο, να επαναληφθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ε, σε εθνικό επίπεδο πιο συγκεκριμένα και επικυροποιημένα δεδομένα. Ε, τι μπορούμε λοιπόν να πούμε, ότι πραγματικά δεν έχουμε εκτιμήσεις τελευταίες, θα πρέπει για να το κατορθώσουμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες μελέτες, χρησιμοποιώντας και μελέτες τηλεμέτρησης. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήσαμε για να μετρήσουμε τα μωρά φώκες βασίστηκαν σε ε, μοντέλα τα οποία, σε πρότυπα αν θέλετε, τα οποία ε, είναι τα ίδια πιστεύουμε, ε, είναι του Ηνωμένου Βασιλείου. Φανταζόμαστε ότι έχουμε παρεμφερεί πληθυσμό αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Πώς έχει τώρα η κατανομή. Από τους διάφορους χάρτες βλέπετε ότι κυρίως μετρήθηκαν οι ακτές οι δυτικές. Άρα έχουμε περιορισμένες πληροφορίες. Όπως σας είπα, γίνονται ε, μετρήσεις ε, τηλεμέτρησης και οποιαδήποτε ε, πρόοδος αυτού του είδους στην τεχνική θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να τα μετρούμε καλύτερα, βεβαίως χρησιμοποιώντας και GPS και GSM θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εικόνα των θηλαστικών τα οποία ζουν στη θάλασσα και να μην έχουμε όλο μετρήσεις αυτών τα οποία φτάνουν στις ακτές. Τι γνωρίζουμε λοιπόν. Ξέρουμε ότι στην Δυτική Εκτή μόνο 17 ε, κοινές φώκες ε, harbor seals, αυτές που φτάνουν στα λιμάνια, έχουν μετρηθεί. Ίσως θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ε, μετρήσεις. Πέρσι όσον αφορά τις ε, γκρίζες φώκες ε, είχαμε 8, είδαμε όμως ότι 4 μετακινήθηκαν προς την Σκοτία για 15 περίπου ε, χιλιόμετρα μετρήθηκαν και μπορούμε να πούμε ότι οι κοινέ ε, ε, φώκες κυνηγούν αν θέλετε και βρίσκονται πιο κοντά στις ακτές οι γκρίζες είναι αυτές οι οποίες βγαίνουν πιο βαθιά στη θάλασσα αλλά θα πρέπει να κάνουμε, όπως σας είπα, περισσότερες ε, ε, μελέτες χρησιμοποιώντας νέες ε, τεχνικές. Τώρα, με τι τρέφονται οι φώκες στην Ιρλανδία. Και πάλι, όπως σας είπα, προσπαθούμε και πάλι να κάνουμε εκτιμήσεις βασιζόμενοι σε μετρήσεις οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ τελευταίες. Όλες οι μελέτες που έχουμε σήμερα είναι απορχαιωμένες, διότι ε, είχαν γίνει την δεκαετία του 1990 και βλέπουμε κυρίως με ποια ψάρια τρέφονται. Πολλά ψάρια και διαφορετικά τρώνε οι φώκες του λιμανιού, κυρίως ε, βυθοπελαγικά. Εδώ βλέπετε ποια είναι τα διαφορετικά είδη ψαριών, ε, γάδο, ρέγγες, βακαλάο, αμόχελα, γενικότερα γαδοειδή. Βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται πολλές φορές και από το βάρος και από το μέγεθος του, ε, της κάθε φώκιας και από το μέγεθος των ψαριών. Εδώ, όπως σας είπα, έχουν γίνει μελέτες και για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και να μας δώσουν στοιχεία έχουμε έρθει ε, σε επαφή με τους ε, διάφορους ε, επαγγελματίες αλληλείς που μας λέγουν ότι οι φώκες τρώνε Εγλεφίνο. και άλλα είδη ψαριών τα οποία βρίσκουν. Έχει βεβαίως αλλάξει η διατροφή τους ανάλογα με τα είδη ψαριών από το 1990 και, τα... και μετά. Υπάρχουν βατραχόψαρα μεταξύ άλλων, άλλο είδη ψαριών και όπως μας είπαν δεν υπάρχει ε, δεν υπάρχουν πάρα πολλά αξιόπιστα στοιχεία, δεν υπάρχει πλήρης ε, ε, κάλυψη, είναι περισσότερο ε, παλιά τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτό το οποίο πολλές φορές ε, καθορίζει τι έχουν φάει είναι τα κεφάλια κάποιων ψαριών που τα βρίσκουν οι ψαράδες στα δίχτυα τους και δεν ξέρουν ε, και καταλαβαίνουν τι ήδη ε, ψάρι έχουν φάει. Μας είπαν επίσης ότι πολλές φορές και βρίσκουν δαγκωμένους σολομού σε κεφάλια σολομού στα δίχτυα τους. Επίσης, όταν ε, δούμε τα αποτελέσματα του, των ειδών διατροφής, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με το τι ε, μέρος του ψαριού, με τι μέρος του ψαριού τρέφονται. Κάτι το οποίο επίσης ε, ε, πρέπει να αναφέρω είναι ότι δεν έχουμε διάφορες, ε, έχουμε λίγες ή σχεδόν καθόλου τεχνικές για να μετρήσουμε αυτό το στοιχείο και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές και συμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Άρα μπορώ να πω ότι δεν έχουμε πολύ καλές εκτιμήσεις και στοιχεία που αφορούν την ε, κατανάλωση ψαριών από τις φώκες στα ύδατα τα Ιρλανδικά και θα πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, μία πολύ μεγάλη και περιστατωμένη ε, μελέτη. Τώρα, η αλληλεία στην Ιρλανδία. Βλέπετε εδώ τα κυριότερα ε, ε λιμάνια, τα κυριότερα είδη, πέλαγικά πελαγικά, ε, αλληλεία ανοιχτή θάλασσα. Πώς επηρεάζεται η αλληλεία τώρα α, κυρίως από τις ε, ε πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε την, ε, την σύγκριση ε, μεταξύ ε, των αλλιευμάτων που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι των αποθεμάτων αλλιευτικών πόρων και την κατανάλωση των, της φώκιας. Δεν έχουμε τέτοιου είδους εκτιμήσεις για την ε, κατανάλωση αλλιευμάτων από τη Φώκια στα Ιρλανδικά ύδατα. Δεν έχουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, τηλεμετρικές ε, τεχνικές που να μας βοηθούν να έχουμε μία σαφή εικόνα. και έχουμε πολύ λίγα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε εκτιμήσεις πιο ε, ακριβείς. Άρα υπάρχουν ανακρίβειες και στα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε. και οι επιπτώσεις της φώκιας στα αλλιευτικά αποθέματα παραμένουν άγνωστες. Τώρα, σε τουρκικό επίπεδο. Έχουμε κάπως περισσότερα στοιχεία χάρη σε μία μελέτη η οποία είχε γίνει, όπως σας είπα, τη δεκαετία, δεκαετία του 90 σε διάφορα αλλιευτικά σκάφη και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε πάρει ε, κυρίως αυτό αφορά την ε, παράκτια αλληλεία εντός 12 ε, μιλίων, τη χρησιμοποίηση ε, τατικών σταθερών διχθείων ή τα ε, σειρώμενα δίκτυα. Ξέρουμε ότι έχουν η τελευταία μέτρηση είναι το 2006, έχουν γίνει αρκετές καταστροφές σε τέτοιου είδους δίχτυα από τις, ε, από τις ε, φώκες. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένους αριθμούς. Έχουμε ε, στοιχεία παλιά, αλλά όχι σημερινά, για να ξέρουμε κατά πόσον η φώκες καταστρέφουν όλα αυτά τα λιευτικά εργαλεία. Τα στοιχεία μας είναι παλιά, της προηγούμενης δεκαετίας. Οι ζημιές όσον αφορά την ε, αλία του Σολομού ε, είναι της τάξεως 1 με 40%. Επίσης έχουμε ε, απώλειες στην ε, υδατοκαλλιέργεια, κυρίως ε, για τον Σολομό, του τάξεως του 20%. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν οι ε, αλληλείς, η Ομοσπονδία Αλλιέων, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένους και πάλι αριθμούς σας λέω. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων. Έχουμε ε, στοιχεία φετινά του 2010. Έχουμε μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα επτά ε, κύρια είδη αλλιευμάτων. Δεν έχουμε πάρα πολύ ε, καλά, σε, καλά στοιχεία για τον ε, Σολομό, τον ε, γάδο και τον βακαλάο μερλάν. Για τον εγλεφίνο πιστεύουμε ότι τα αποθέματα είναι καλύτερα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μικρή ε, αύξηση. Εδώ σε αυτό τον πίνακα έχετε ανάλογα με τα χρώματα που βλέπετε την ε, κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων στα ύδατα της Ιρλανδίας και ανάλογα με τα χρώματα, την περιοχή και το είδος βλέπετε την εκτίμηση όσον αφορά τα αποθέματα καθώς και τις ε, ε συμβουλές που δίδονται για να μπορέσουν να ε, διατηρηθούν ή να βελτιωθούν τα αποθέματα. Δεν έχουμε, όπως βλέπετε, όμως συγκεκριμένους αριθμούς. Δεν μπορούμε ούτε καν να μετρήσουμε την, ε, τον ανταγωνιστικό. Ξέρουμε όμως ότι ε, προκαλούν οι φώκες αρκετά ε, μεγάλα προβλήματα. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις και τα παρεπιμ, στα παρεπιμπτωτά αλλιεύματα. Δηλαδή, ποια είναι τώρα η επίπτωση της αλίας, της φώκες. Ε, υπάρχουν τέτοιου είδους παρεπίπτοντα αλλιεύματα, δεν έχουμε όμως ε, συγκεκριμένα ε, αριθμούς. Κυρίως οι φώκες που πιάνονται τα δίχτυα είναι μικρές σε διάσταση, είναι τα μωρά. Βεβαίως θα πρέπει πάντα να ε, μετρώνται αυτά τα παρεπίμπτωνα αλλιεύματα. Θα πρέπει να ξέρουμε σύμφωνα με κάποια μελέτη που πρέπει να γίνει ποιος είναι ο αριθμός τους και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει κάποια μελέτη. Είναι σημαντικό να πιάνονται ε, ζωντανά και τα, τα μικρά της φώκες και να δίδονται και για μελέτες. μέτρα ελέγχου των ε, αρπακτικών Πρέπει να υπάρχουν μέτρα ως αναφορά και τον, ε, τα όπλα που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο θανατώνονται οι φώκες. Χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα, διάφορες ε, ε, τεχνικές για να αποτραπούν οι φώκες, χρησιμοποιούνται διάφορα ε, πομπή ε, που εκπέμπουν ακουστικά ε, ηχητικά μηνύματα. Ε, και βεβαίως κανένας μέχρι τώρα δεν έχει ε, προσέξει στη δικαιοσύνη όλους αυτούς τους ε, λαθροκυνηγούς, όλους αυτούς οι οποίοι θανατώνουν τα μωρά της φώκιας. Τέτοιου είδους προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν να προστατευτεί η αλληλή, αλλά βεβαίως δεν θα πρέπει να θανατώνονται και με άγριο τρόπο τα μωρά φώκιας. συμπεραίνοντας θα πω ότι πραγματικά δεν ε, γνωρίζουμε ποιο είναι το ε, επίπεδο ε, βιολογικού ανταγωνισμού και διάδρασης μεταξύ αλληλείας και φώκιας στα υδατά μας. Θα πρέπει να γίνουν ειδικέ μελέτες. Προς το παρόν, οποιαδήποτε μέτρα έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν ήταν αποτελεσματικά και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, μελέτες πιο συγκεκριμένες για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια κενά και να έχουμε περισσότερη γνώση του όλου προβλήματος. Και βεβαίως θα χρειαστούμε χρόνο να εφαρμόσουμε τέτοιες τεχνικές, αλλά θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες όσο δεν, αυτές, όσο δεν έχουν γίνει αυτές οι μελέτες και οι έρευνες από τον, σε επαγγελματίε, από τους αλληλείς και φαντάζομαι ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν για να κάνουν τέτοιους μελέτες. Ε, στις αρχές του 90 Δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας από όλου του ενδιαφερόμενους για να κάνει τέτοιου μελέτες, αλλά λίγα χρόνια μετά ε, διαλύθηκε και έτσι δεν έχουμε βρει ακόμη τις κατάλληλες λύσεις. Αυτό το οποίο προτείνουμε λοιπόν είναι να θεσπιθεί στη μια ομάδα διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο ε, με την συμμετοχή, όπως σας λέω, όλων των ενδιαφερομένων από την ε, αλληλεία, ε, από κυβερνητικούς εκπροσώπους, από πανεπιστημιακούς για να μπορέσουν να γίνουν οι σωστές μελέτες και οι σωστές μετρήσεις για να δούμε ποια είναι τα αποθέματα και αλληλευτικά και οι επιπτώσεις της φώκιας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κρόνιν. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τα δεδομένα αυτά και να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε με τη Σκοτία. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χάκαν Βέστερμπεργκ από το Σουηδικό Συμβούλιο Αλίας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την αρνητική αυτή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις φώκες και τα αλληλευτικά αποθέματα. Τον καλωσορίζω λοιπόν και του δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση θα μιλήσω για κάποιες ε, διαχειριστικές λύσεις. Όσον αφορά την ε, διένεξη αυτή, την αρνητική ελληνεπίδραση ανάμεσα στις φώκες και τα από αποθέματα. Θα ξεκινήσω με μία σύντομη συζήτηση της φύσης της διένεξης αυτής και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε κάποιες μεθόδους ε, τεχνικού μετριασμού. Επίσης θα μιλήσουμε για κάποια συστήματα οικονομικής αντιστάθμισης, για το προστατευτικό κυνήγι, για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων. Και στο τέλος θα αναφερθώ στις καλύτερες δυνατέ μεθόδους που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε για το μέλλον. Ας μιλήσουμε όμως καταρχάς για τη φύση της ε, σύγκρουσης, τη διένεξή αυτή. Δεν υπάρχει μία μόνο τέτοια διένεξη, αρνητική αλληλεπίδραση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαστάσεις που έχουν να κάνουν με το είδο της φώκια και με το είδο των ελευτικών αποθεμάτων. Θα λέγαμε επίσης ότι η σύγκρουση αυτή είναι αμοιβαία. Από τη μία πλευρά δηλαδή και από την άλλη υπάρχει αρνητική αλληλεπίδραση. Από την αλία προς τις φώκες και από τις φώκες προς την αλία. Στην γραφική αυτή παράσταση βλέπετε τις δύο διαφορετικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η διένεξη αυτή. Καταρχάς βλέπετε το γεωγραφικό πλάτος. Περισσότερες φώκες έχουμε στο βορρά Η ε, αλληλεπίδραση λοιπόν η αρνητική εκεί και ο ανταγωνισμός αυξάνεται στο βορρά. Και η άλλη διάσταση είναι η αλία. Από τη μια έχουμε την ε, αλία, την παρακτια μικρής κλίμακος και από την άλλη έχουμε την αλία που γίνεται στα νυχτά και είναι μια αλία μεγάλης κλίμακος. Και η μεγαλύτερη αρνητική αλληλεπίδραση εντοπίζεται κυρίως στην ε, παράκτια μικρή αλία τόσο στις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα λιεύματα και στα εργαλεία και όσον αφορά την παρεπίμπτουσα σαλία. Και σαφώς υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τη διατήρηση, την προστασία των ειδών, ιδίως όταν εντείνεται η σύγκρουση αυτή ανάμεσα στα δύο είδη. Ας περάσουμε τώρα σε μεθόδους ε, μετριασμού της σύγκρουσης αυτής. Ποια είναι τα τεχνικά μέσα που έχουμε στη θέση μας. Βλέπουμε καταρχάς ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε τα αλλιευτικά εργαλεία, προκειμένου αυτά να μην πλήττονται τόσο πολύ από τις φώκες, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να μετεγκαταστήσουμε και τις ε, φώκες ή να χρησιμοποιήσουμε και άλλους μηχανισμούς εκφοβισμού των φωκών. Για την προστασία των ε, αλλιευμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέες παγίδες ψαριών ή ηχθειοφραγμούς, τουλάχιστον να μετατρέψουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία εκτίθονται όλο και περισσότερο σε ζημιές από τις φώκες. Αν θέλετε, πρόκειται για τις πιο παραδοσιακές μεθόδους αλίες που χρησιμοποιούνται από πάρα πολύ παλιά και ακόμα χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Να φέρομαι στις παγίδες ψαριών και στους ηχθειοφραγμούς. Μία λύση λοιπόν θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα πιο ισχυρό υλικό στα δίκτυα. Ένα υλικό δηλαδή που δεν θα επέτρεπε στα μάλλον στις φώκες να καταστρέψουν τα εργαλεία και να έχουν πρόσβαση στα ψάρια. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν νέα δίκτυα, νέο κυκλίδωμα μεταλλικό στις ε, παγίδες. Βλέπετε εδώ πέρα ένα παράδειγμα για μια λύση που είχε χρησιμοποιηθεί στη Βαλτική θάλασσα, όπου έχουμε κυρίως, ελία Σολομού. Χρησιμοποιείται εδώ πέρα πολύ μεγάλη κλωβή, η οποία είναι γυροβολημένη στην ακτή και απέχουν περίπου 500 μέτρα από την ακτή και επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Βλέπετε εδώ πέρα μια φωτογραφία που έχει βγει από τον κλωβό προς τα δίχτυα εκείνα που κρατά τον κλωβό αγκυροβολημένο. Η λύση λοιπόν που έχει προβλεφθεί για τη χρησιμοποίηση αυτού του εργαλείου είναι το εργαλείο αυτό να γίνει πιο φιλικό προς το χρήστη και να είναι πιο αθεκτικό στις ζημιές από τις φώκες. Έχετε εδώ πέρα κάποιες σχεδίες, φουσκωτές σχεδίες, οι οποίες ε, συνήθως βρίσκονται μέσα στο νερό, μέσα στο βυθό. Αρχίστε σιγά σιγά να φουσκώνετε τις σχεδίες αυτές, αυτές φουσκώνοντας ανεβαίνουν προς την επιφάνεια και κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διάσετε τα αλλιεύματα μέσα στο σκάφος σας. Και στη συνέχεια στην άλλη φωτογραφία βλέπετε την τελική είσοδο μέσα στον ε, κλωβό και έχει ένα πλέγμα είσοδος αυτή, το οποίο προστατεύει το εργαλείο αυτό από τη φώκια. Η φώκια προφανώς δεν μπορεί να μπει μέσα στο θάλαμο αυτό το μεταλλικό. Το πρόβλημα όμως που προέκυψε είναι ότι οι κυφώκες άλλαξαν συμπεριφορά. Αντί να προσπαθούν να μπουν μέσα στον κλοβό, περιμένουν έξω από τον κλοβό και προσπαθούν να πιάσουν τα ψάρια τη στιγμή που μπαίνουν μέσα στον κλοβό. Βλέπετε εδώ πέρα μια γραφική παράσταση που δείχνει την ε, πορεία της φώκιας αλλά και την πορεία των αλλιέων κατά την αλία Σολομού Βλέπετε εδώ πέρα η φώκια περιμένει έξω από την παγίδα και ξαφνικά πετάγεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να καταφέρει να πάρει τα λιεύματα. Για να λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό, χρειάστηκε να επανασχεδιάσουμε και το ίδιο το τμήμα αυτό της ε, εισόδου προς την παγίδα αυτή, προκειμένου να αποφύγουμε όλες τις έντονες γωνίες ε, που θα βοηθούσαν ουσιαστικά τις φώκες να πιάσουν τα ψάρια που μπορεί να είχαν κολλήσει εκεί και θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης δίχτυα ένα κυκλίδωμα με ε, μεγάλο μάτι, με μεγάλο βρόχο προκειμένου να μπορούν να περνάνε μέσα από αυτό τα ψάρια. Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα αποθαρρύνουμε τις φώκες ακόμα και στη νέα αυτή συμπεριφορά που έχουμε υιοθετήσει. Που έχουν υιοθετήσει, με συγχωρείτε. Έχουμε λοιπόν ένα νέο θάλαμο, μια νέα παγίδα, καθώς επίσης και ένα νέο σχεδιασμό του Και χρησιμοποιείται πλέον το νέο αυτό σύστημα σε πάρα πολλές γεωγραφικές ε, ζώνες, κυρίως στην Βαλτική. Και ο νέος αυτός σχεδιασμός, η νέα παγίδα, μας επιτρέπει να προσθέσουμε πολύ περισσότερο τα λιεύματα Σολομού. Τα άλλα αληφτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε είναι τα στάσιμα πλάδια. Και αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις φώκες και είναι και πιο δύσκολα ακόμα να τα προστατεύσουμε. Η εναλλακτική μέθοδος λοιπόν, την οποία έχουμε επινοήσει, είναι η χρησιμοποίηση μιας άλλης αλληλευτικής μεθόδου πολύ απλά. Οι εναλλακτικέ λοιπόν ποιες είναι, κυρίως η αλία με η χρησιμοποίηση κιούρτου. Στα πλαίσια της αλίας της Βαλτικής τα στάσιμα απλάδια χρησιμοποιούνται πολύ για την αλίευση γάδου, ένα περίπου ίμιση, το 50% της συνολικής αλίευσης γάδου γίνεται με στάσιμα απλάδια. αλλά η μέθοδος αυτή δυσχεραίνει πάρα πολύ εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφοράς των φωκών. Στην κεντρική Βαλτική, για παράδειγμα, ένα 80% των αλλιευμάτων καταστρέφεται από τις φώκες, όπου χρησιμοποιούνται ιδίω ε, στάσιμα απλάδια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την αλίευση, τουλάχιστον με αυτή την αλλιευτική μέθοδο. Αυτό που ξεκινήσαμε λοιπόν να επεξεργαζόμαστε είναι να χρησιμοποιείται ένας επιφανειακός σκιούρτος για την ε, Αλία Σολομού. Ο κιούρτος αυτός βρίσκεται ορισμένα μέτρα πάνω από, την, ε, από το βυθό της θάλασσας. Είναι εγκυροβολημένος δηλαδή, ενώ βρίσκεται ακόμα μέσα στη θάλασσα μπορεί ο Σολομός να μπει μέσα στον κιούρτο αυτό και στη συνέχεια οδεύει προς τα πάνω και εκεί πέρα παγιδεύεται, στο ανώτερο τμήμα δηλαδή του κιούρτου. Και από ό,τι φαίνεται η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συναλλακτική, παρουσιάζει πολλές δυνατότητες, αλλά θα πρέπει να επεξεργαστούν περισσότερο τις λεπτομέρειες της μεθόδου αυτής, και θα πρέπει το εργαλείο αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό. Πάντως παρουσιάζει τα ίδια πλεονεκτήματα με τα στάσιμα απλάδια. Αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από μικρούς αλείς, δεν απαιτείται δηλαδή ένας σημαντικός εξοπλισμός και η ποιότητα των ελευμάτων παραμένει υψηλή ποιες μεθόδους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκφοβήσουμε τώρα τις φώκες. Χρησιμοποιούμε κάποιες συσκευές ακουστικής παρενόχλησης AHD που έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως από εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. Στις εγκαταστάσεις αυτές, αυτές οι συσκευές μπορούν όντως να αποδειχθούν αποτελεσματικές. Είναι πολύ δύσκολο όμως να χρησιμοποιηθούν οι συσκευές αυτές σε άλλες μεθόδους αλίας, γιατί χρησιμοποιούν πολύ ηλεκτρική ενέργεια και καταλαβαίνετε ότι ε, η ηλεκτρική αυτή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, ιδίως σε ένα μικρό λευτικό σκάφος. σε μικρά επίπεδα ηλεκτρικής ενέργειας ε, λειτουργούν διαφορετικά και ουσιαστικά έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Καλούν τις φώκες να έρθουν προς το σημείο αυτό για να τραφούν. Ποιες άλλες μεθόδους έχουμε δοκιμάσει. Η μετεγκατάσταση είναι μία μέθοδος. Έχει χρησιμοποιηθεί στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και αποδείχτηκε τελικά ότι οι φώκες επιστρέφουν, καταφέρουν να καλύψουν πολύ γρήγορα μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις, επομένως δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η μέθοδος αυτή της μετεγκατάστασης. Επίσης, Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η αποτροπή της φώκιας με διάφορες μεθόδους. Ξέρετε για παράδειγμα ότι αν δηλητηριαστείτε μια φορά δεν θα ξαναφάτε το ίδιο φαγητό πολύ ευχάριστα την επόμενη φορά. Η μέθοδος αυτή της δηλητηρίασης ε, χρησιμοποιείται στις ε, φώκες. Όλα τα θηλαστικά αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή για τους λύκους. Για κάποια μεγάλα αρπακτικά. Αλλά είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί η μέθοδο της δηλητηρίασης στις φώκες. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολύ καλά ποια φώκια τρώει τελικά το δηλητηριασμένο αυτό φαγητό, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λίγο ακόμα τη μέθοδο αυτή και να την παρακολουθήσουμε καλύτερα. Ενδεχομένως να υπάρχουν και νέες δυνατότητες που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει. Μία άλλη μέθοδος είναι να κρύψουμε τα αλλιευτικά εργαλεία. Αν για παράδειγμα η φώκια δεν είναι σε θέση να εντοπίσει μια σημαδούρα που βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, ενδεχομένως να μην έρθει προς το σημείο αυτό που βρίσκω τελευταία από θέματα, αλλά ακόμα και η μέθοδος αυτή της απόκρυψης δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Μία πτυχή, αν θέλετε, του όλου προβλήματος είναι και η παραπίπτουσα αλία. Πολύ συχνά δηλαδή οι αλληλείς εγκαταλείπουν τα αλληλευτικά εργαλεία μέσα στη θάλασσα μετά την αλληλευτική προσπάθεια. Πάνω σε αυτά έχουν πιαστεί και άλλα αλλιεύματα τα οποία δεν επιθυμούν οι αλληλείς και καταλαβαίνετε ότι και αυτό με τη σειρά του συμβάλλει καθότι προσελκύει τις φώκες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μειωθεί η του Τώρα, το ζήτημα της οικονομικής ε, αποζημίωσης, οικονομικής αντιστάθμισης. Καταρχάς πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αντιστάθμιση για τις ζημιές που έχουν ε, προκληθεί, πόσο μάλλον από είδη τα οποία προστατεύονται. Από ό,τι φαίνεται τελικά ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού είναι υπεύθυνο για το συνολικό κόστος της ε, διατήρησης και της προστασίας που αποφασίζει μια μεγάλη πλειονότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικής αλληλεπίδρασης στο ζωικό βασίλειο έχει συστηθεί το ζήτημα αυτό και στην περίπτωση της, ΦΟΚΕΣ έχουμε λάβει υπόψη μας και τις ε, κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι θα μπορούσαν να επιτραπούν τέτοιες επιδοτήσεις, τέτοιες ενισχύσεις, αλλά δεν έχει δώσει την απόλυτη έγκρισή της. Έχει ακόμα μια σκεπτικιστική στάση. Η οικονομική αποζημίωση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την αλία μικρής κλίμακος. Θα επέτρεπε στην αλία αυτή να επιζήσει μέχρι να βρεθεί μία πιο μόνιμη λύση, μία πιο μόνιμη τεχνική λύση μετριασμού. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έπρεπε να διονυστεί μια τέτοια επιδότηση, γιατί θα γινόταν τελικά αντιαποτελεσματική. Α περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει πάλι με το ζήτημα αυτό της διένεξη ανάμεσα στις φώκες και λευτικά αποθέματα και πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα του κυνηγιού, κυνήγι φώκες. Υπάρχουν εδώ πέρα δύο επίπεδα σε αυτό το κυνήγι. Το προστατευτικό κυνήγι, όπου χορηγούνται ειδικέ άδειε κυνηγιού για τοπικά σχέδια μετριασμού και τα σχέδια αυτά χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις χώρες στις οποίες παρατηρείται αρνητική ελεπίδραση ανάμεσα στις φώκες και τα λεφτικά αποθέματα. Οι αλληλείς δηλαδή έχουν άδειε κυνηγιού φώκιας και η βασική ιδέα εδώ είναι να ε, γίνει μία μείωση του πληθυσμού των φωκών εκείνων που συμβάλλουν περισσότερο στη μείωση των ελευτικών αποθεμάτων. Επίσης ε, προβλέπεται σε ορισμένες περιοχές μία περίοδος ε, κατά την οποία επιτρέπεται το κυνήγι της φώκιας και μάλιστα με μια συγκεκριμένη περιορισμένη ποσόστοση. Κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, συμβαίνει στη Βαλτική. Λειτουργεί το σύστημα αυτό πάντως. Ελάχιστες αξιολογήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα αυτών των αδειών για το περιορισμένο κυνήγι φώκες. Στη Σουηδία το κυνήγι απαγορεύτηκε εντελώς για 20 περίπου χρόνια και στη συνέχεια το 1900 90, περίπου πριν από 10 χρόνια. Ξεκίνησε μια δοκιμή, ουσιαστικά προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων της ε, χρησιμοποιούμενης μεθόδου. Δηλαδή, σε μια συγκεκριμένη περιοχή προσπαθήσαμε να αποτιμήσουμε την ε, ζημιά που έχει γίνει στα λιευτικά εργαλεία και στα λιευτικά αποθέματα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη περιοχή ελέγχου 50 χιλιόμετρα μακριά στη συνέχεια, όπου γινόταν πάλι μια αντίστοιχη αποτίμηση και παρακολούθηση των ζημιών. Και στη συνέχεια σκοτώθηκε ένα συγκεκριμένο αριθμό φωκών πάλι σε κάποιε περιοχέ όπου κάναμε πειράματα και προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα ανάμεσα στι περιοχέ εκείνε όπου είχε μειωθεί με του φεκισμό ο πληθυσμό τη φώκια και στι υπόλοιπε. Στη μία περίπτωση βλέπετε ότι οι ζημιές συνέχισαν να αυξάνονται Ακόμα και εκεί που ε, είχαμε κυνηγήσει τις φώκες, βλέπετε εδώ πέρα τον αριθμό των φωκών που σκοτώθηκαν. Για μια περίοδο δύο εβδομάδων περίπου έγινε το κυνήγι αυτό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι ζημιές. Συνεχίζονται και μετά το τέλος της περίοδου του κυνηγιού και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο. Βλέπετε λοιπόν τα αποτελέσματα πριν και μετά την περίοδο κυνηγιού. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ε, όσον αφορά τις rough seals, το είδος αυτό, υπήρξε μία επίπτωση. Χωρίς όμως αυτή να είναι πάρα πολύ σημαντική, τουλάχιστον για την, περίοδο της, για την περιοχή της Βαλτικής. Η σημαντικότερη επίπτωση όμως που έχετε είναι μια ψυχολογική επίπτωση αν θέλετε. Ψυχολογική επίπτωση για τους αλλείς. Έχουν ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο ένα δικαίωμα αυτοάμυνας. Είναι σημαντικό ένας ψαράς να νιώθει ότι μπορεί να προστατεύσει την παραγωγή του. Έχουμε πίτα και το δεύτερο επίπεδο κυνηγιού όπου έχετε το δικαίωμα να κυνηγήσετε μία ρυθμισμένη ε, ένα ρυθμισμένο πληθυσμό φώκιας, δηλαδή ένας, ε, έχουμε ένα, μια ρυθμισμενη ενα ρυθμισμενο πληθυσμο φωκιας δηλαδη εχουμε ενα μια μειωση του πληθυσμού η οποία είναι προαποφασισμένη. Έχει ως στόχο να κρατήσει τον πληθυσμό σταθερό. Και πάλι όμως εδώ πέρα βλέπουμε ότι η επίπτωση δεν είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί τελικά η κατανάλωση ψαριών που γίνεται από τις φώκες δεν είναι τόσο σημαντική σε σχέση με άλλα είδη όπως τα κοιτοειδή. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες περιοχές και για συγκεκριμένα ψάρια η θύρευση από τις φώκες μπορεί να είναι σημαντική και εκεί πέρα το ελεγχόμενο αυτό κυνήγι μπορεί να αποβεί αποτελεσματικό. Και πάλι όμως είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε σφαιρικά τη μέθοδο αυτή. Και ακόμα και το να εντοπίσουμε κάποιες επιπτώσεις, οι επιπτώσεις αυτές δεν θα είναι απαραίτητα ευνοϊκές, δηλαδή δεν θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε μείωση της ε, κατανάλωση λευτικών αποθεμάτων από τις φώκες μπορεί να έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε ότι αν ε, εξαφανίσουμε τις ε, φώκε, αυτόν τον θηρευτή δηλαδή, μπορεί να εμφανιστεί ένας άλλος θηρευτή, ένα άλλο ενδιάμεσο αρπακτικό, το οποίο μπορεί και αυτό με τη σειρά του να καταναλώνει λευτικά αποθέματα και μάλιστα μπορεί να έχει ακόμα και πιο επιζήμιες επιπτώσεις. Πάντως, Βλέπουμε ότι η κατάσταση παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με βάση την κάθε τοπική περιοχή και το κάθε είδος ψαριού. Επομένως, ε, απαιτείται μία σφαιρική εις βάθος ανάλυση κατά περίπτωση για κάθε είδος και κάθε γεωγραφική περιοχή. Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να διαχωρίσουμε να, να επιλύσουμε το πρόβλημα διαχωρίζοντας τις περιοχές στις οποίες γίνεται τελεία και στις οποίες ζουν οι φώκες. <laughs> Αυτό βέβαια δεν ε, έγινε, δεν εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό ο καθορισμός ε, προστατεμένων ζωνών ε, δεν ε, ε, έγινε αρκετά ευρέως τους ώστε να επηρεάσει την σύγκρουση αν θέλετε αλίας και ε, φώκιας. Το τελικό μήνυμα λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία. Ποιο είναι. Έχουμε κάποια στοιχεία για τη διατροφή της φώκιας, για τους πληθυσμούς της φώκιας, για το επίπεδο σύγκρουση και τα λοιπά, αλλά δεν αρκούν. Θέλουμε και άλλα στοιχεία και άλλες πληροφορίες. Πρέπει να εσλεχθούν αυτές κατά προτεραιότητα. Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι επιστήμονες είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα αυτό και επιστημονικές μέθοδοι Συγγνώμη, δεν είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι εδώ και οι επιστημονικές μέθοδοι δεν ξέρουμε εάν θα μπορέσουν να επιλύσουν ε, από μόνες τους τη σύγκρουση αυτή. Υπάρχουν και κοινωνικές πτυχές γιατί ε, υπάρχουν ολοκλήρες κοινωνίες ε, αλλιέων σε ορισμένε περιοχές υπάρχουν και άλλες πτυχές στην όλη υπόθεση πρέπει κανείς να βρει λύσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους διάφορους είναι σημαντικό αυτό Εμείς καταφέραμε στη Σουηδία να κάνουμε κάποια πράγματα και να είμαστε σχετικά επιτυχείς ιδιαίτερα σε σχέση με μεθόδους που δεν σκοτώνουν μετρίασης ε, που δεν σκοτώνουν μετριασμού με συγχωρείτε που δεν σκοτώνουν τελικά τις ε, φώκες είχαμε καλά αποτελέσματα εκεί αλλά είναι επίσης σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αφού ο πληθυσμός των φωκών α, δεν είναι σταθερός και η σύγκρουση δεν είναι σταθερή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο πληθυσμός της γκρίζας φωκιάς στη σκοτία παλιά ήταν ασήμαντος ε, και σε 20 χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικός. Η διαχείριση λοιπόν θα πρέπει και αυτή να προσαρμοστεί στο, στον πληθυσμό που κυμαίνεται, που αυξάνεται, που μειώνεται για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Οι μέθοδοι μετριασμού θα πρέπει να προσαρμόζονται και αυτές και για το, όσον αφορά τον πληθυσμό της φώκης αλλά και όσον αφορά την αλληλευτική, τις αλληλευτικές δραστηριότητες. We've heard the four Ακούσαμε λοιπόν όλες τις παρουσιάσεις που ε, περιέργως μας ε, ε, δείχνουν ότι άλλα αρπακτικά ψάρια ή θαλασσοπούλια είναι πιο επικίνδυνα τελικά για τα λευτικά αποθέματα από ότι οι φώκες. Επίσης, από όλους ακούσαμε αυτό που ότι αν ακόμη και να αφαιρέσουμε αν θέλετε από κάποια οικοσυστήματα όλες τις φώκες αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα αλλιευτικά αποθέματα. Αυτό είναι εκπληκτικό σαν συμπέρασμα, σαν μήνυμα αν θέλετε που βγαίνει από όλες αυτές τις παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό στους αλληλείς της ε, Δυτικής Σκοτίας. Ε, δεν νομίζω ότι θα το καλοδεχτούν το μήνυμα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ας ε, αρχίσουμε τη συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο, κύριος Χάγκλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τέσσερις ε, εμπειρογνώμονες που μόλις έκαναν τις παρουσιάσεις τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνουμε σήμερα την ακρόαση αυτή γιατί ε, ε το θέμα που κουβεντιάζουμε με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Προέρχομαι από τη Φινλανδία βεβαίως, αλλά ε, δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τη Φινλανδία, αλλά για ολόκληρη τη Βαλτική. Στη χώρα μου χάσαμε το 50% των αλλιέων μας τα τελευταία χρόνια η Φώκια και η Κορμοράνη και ο Κορμοράνος είναι ο κυρίως λόγος για τον οποίο χάνουμε αν θέλετε τους αλληλείς μας και μειώνεται τόσο σημαντικά η ελευτική δραστηριότητα των συμπολιτών μου η κύρια τα λευκά είδη ψαριού και ε, τους σολομούς καταναλώνουν οι φώκες και τα οι ποσότητες αυτών των ειδών που που τρώνε οι φώκες ε, κατά την δική μας άποψη και βάσει των μελετών που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αλλιεύονται. Γι' αυτό εκπλήσωμαι που άκουσα από τους ομιλητές να λένε ότι αναφερούσαμε τις φώκες από το οικοσύστημα δεν επηρεαζόταν τα πράγματα. Λάθος κατά τις δικές, κατά τις δικές μας μελέτες, τουλάχιστον ειδικά για τη Βαλτική, επειδή και ίσως και ο πληθυσμός της Φώκιας αυξάνεται ε, ταχύτατα, ε, τα πράγματα είναι... Ε, διαφορετικά επηρεάζονται, σημαντικά και πολύ αρνητικά η αλλιευτική δραστηριότητα, η αλλία Δε, εκτός αν κατάλαβα λάθος αυτά που είπατε, η εντύπωσή μας στην ε, Φινλανδία είναι τελείως διαφορετική. Ο πληθυσμός, το εισφόκια στην ε, Φινλανδία αυξάνεται συνεχώς και άρα και οι ζημιές στην αλία αυξάνονται όσον αφορά το, το κυνήγι της ε, δεν αποδίδει ε, η μέθοδος αυτή εκτός βέβαια αν αρχίσετε να κυνηγάτε το χειμώνα που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα Βεβαίω εκτός του κυνηγιού δεν υπάρχουν και πολλές άλλες εναλλακτικέ λύσεις η ανάγκη ανάπτυξη νέων αλληλευτικών μεθόδων και εργαλείων μπορεί να βοηθήσει βεβαίως αλλά μέχρι στιγμής ε, δεν ε, ε, βλέπουμε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα εκτός βέβαια αν τρώτε μονίμως νορβηγικό σολομό και όχι φινλανδικό σολομό η κατάσταση στη Φινλανδία είναι κακή πρόεδρος θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μετά αφού γίνουν κάποιες ερωτήσεις η κυρία Λόβακ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 Eh, vill eh, Det var väldigt... Eh, Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν, πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ ενημερωτικές και όπως ήδη ελέγχθη περιέρχως συμφωνούν, συμφώνησαν όλοι οι ομιλητές ότι βεβαίως ε, δεν ε, υπάρχουν ποσοτικοί, δεν μπορούμε να εκφράσουμε ποσοτικά τα αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα για την αλληλεία, αλλά είναι, μας είπαν, πολύ μικρές οι ζημιές τελικά στην αλληλεία. Ε, τα άκουσα όλα αυτά, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Ο πληθυσμό της Φώκιας συνεχώς αυξάνεται. Βεβαίως και η άλλες περιβαλλοντικές απειλές συνεχώς αυξάνονται ε, για δηλητηρίαση ε, υπάρχουν δύο ε, ε, έχουμε πολύ περισσότερες διοξίνες στο περιβάλλον που ε, ε, ε παραμένουν, αποθηκεύονται τρόπον την, στο λίπος ε, και οι διοξίνες αυξάνονται όλο και περισσότερα. Από εκεί πέρα υπάρχουν απειλές και για τα μικρά, για τα νεογνά, διότι στις βόρειες ιδιαίτερα περιοχές ε, στις στις πολικές περιοχές ε, όπου γεννιούνται τα νεογνά υπήρξαν είδαμε ότι πρόσφατα συνέφησαν πολλά πράγματα που επηρέασαν τα νέα αυτά άτομα και πρόσφατα διάβασα μια μελέτη για το πόσο πλήττονται οι πληθυσμοί της α, ακόμη και σε πολύ μικρή ηλικία στις περιοχές αυτές. Θέλω να πω ότι οι πληθυσμοί της Φώκιας απειλούνται από πάρα πολλές αιτίε πέρα από το κυνήγι της Φώκιας από τους σαλίες Ε, θα με ενδιαφέρε να ακούσω ποια είναι, ποιοι ήταν οι πληθυσμοί της Φώκιας πριν από 100 χρόνια σε σχέση με τους σημερινού πληθυσμούς. Από ό,τι γνωρίζω, δεν θυμάμαι, μας είπατε τώρα ότι κάποιο είδος φώκιας ας πούμε σήμερα είναι 20.000 αλλά νομίζω ότι στις αρχές του αιώνα συνολικά α, ναι, ο πληθυσμό ήταν ε, μεγαλύτερο και ο συνολικό πληθυσμό για όλα τα είδη φόκια ήταν 300.000 άτομα. Α, δεν ξέρω αν είναι σωστά τα στοιχεία αυτά. Αυτή τη στιγμή, αν τα στοιχεία μου είναι σωστά, ε, σήμερα ε, έχει επιβιώσει μόνο το 10% των θαλάσσιων θηλαστικών σε σχέση με το αντάτομα που υπήρχαν πριν από 100 χρόνια στο ε, συζήτησα με εμπειρογνώμονες και με τον φίλο Γαρκόνεν του Μουσείου ε, της ε, Σουηδικού Μουσείου ε, και συζήτησα το πάχος το, το πάχος του λίπους ε, των ε, θηλαστικών αυτών το οποίο συνεχώς μειώνεται η μείωση όμως του λίπους του, ε, στα ζώα αυτά είναι κάτι το αρνητικό για την υγεία τους θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε στοιχεία και γι' αυτό το, για αυτή την πτυχή. Δεν ξέρω οι Άισες τι μελέτες έχει ε, κάνει σχετικά και δεν θέλει και μερικά στοιχεία για το πώς αναπτύσσονται τα αποθέματα φώκιας πλέον και αν ε, πλησιάζουν ένα κάποιο σημείο σταθεροποίηση γιατί για κάποια είδη φώκες νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ε, σταθεροποίησης δεν θα σας κουράσω περισσότερο θα πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η, σημερινή ακρόαση κατά την άποψή μου και οι παρουσιάσει πολύ ενδιαφέρουσε για το κυνήγι της φώκια και το, το φεκισμό, το πυροβολισμό της φώκια, να πω ότι φτιάχτηκε μια ταινία όπου, που γυρίστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές και άμα δει κανείς τα ε, το φιλμ αυτό συνειδητοποιεί ε, πώς επιβιώνει αν θέλετε το είδος αυτό για το οποίο μιλούμε γιατί από 100 ε, άτομα ας πούμε μόνο 10 τα 110 άτομα ήταν ιδιαίτερα ικανά για να ξεπεράσουν για να γλιτώσουν και από αυτά τα 10 ιδιαίτερα ικανά άτομα υπήρχαν τρία μονάχα που επιβίωσαν στο τέλος ε, είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να, να δούμε δούμε και πώς επιβιώνει το είδος, αν θέλετε. I think it was Mr. Harkonnen who said that... Σας ευχαριστώ, είπε ο κύριος Harkonnen ότι στα φιόρδες της ε, σκανδιναβικές χώρες το κυνήγι ε, της ε, φώκιας ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι στα, στη Σκοτία και είχε επιπτώσεις τα λέμε. Ίσως θα μπορούσε να επαναλάβει ο συνάδελφος σχολείου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ο κύριος Γκάλαχερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητέ που μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πρέπει να πω ότι με εκπλήσει το ότι μόνο το 1% των ε, ε, αλλιευτικών αποθεμάτων σημαντικών ε, ειδών ε, αλλιευμάτων επηρεάζεται από την φάλα, να με εμποσιάζει αυτό. Συγγνώμη, τη φώκια. Uh, Βεβαίως, θα μπορούσα να επικρίνω την ε, χώρα μου δια το τι uh, ακριβώς κάνει όσον αφορά ε, τις φώκες. Είδα πραγματικά πόσες λίγες υπάρχουν, πόσο λίγες φώκες, οι γκρι, οι φώκες του λιμανιού στην Ιρλανδία και νομίζω ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μελέτες ώστε να γίνουν ε, εκτιμήσεις. Φαντάζομαι ότι καμία χώρα δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό από μόνη της. Θα πρέπει και να τεθούν πόροι από κοινού και να μοιραστούμε όλοι τα πορίσματα των ερευνών. Το θέμα βέβαια της ε, ε διατροφής τους επίσης είναι σημαντικό. Τι, το τι είδος ε, πελαγικά ε, είδη αλίας καταναλώνουν επίσης είναι σημαντικό. Και βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποια είδη, με την ρέγγα, με κάποια άλλα είδη τα οποία πρέπει να προστατεύονται, τα οποία δεν πρέπει να αλλιεύονται, αλλά βλέπουμε ότι καταστρέφονται έξω. Επί, τελειώνοντας τελευταία την λεπτομέρειες, ήθελα να πω ότι ήταν ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις. Αυτό που με απασχολεί επίσης είναι το θέμα της καλλιέργειας που είναι ένα είδος καλλιέργεια που πρέπει να προστατεύσουμε και σήμερα βλέπω ότι απειλούνται ε, από τις φώκες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε και όλοι στις χώρες μας θα πρέπει σε συνεργασία με τα Υπουργεία μας και με την Κομισιόν να κάνουμε μία εμπεριστατωμένη και σφαιρική εκτίμηση της όλης κατάστασης. Και έχοντας ακούσει σήμερα τι ελέγχθη, έχω την εντύπωση ε, ότι καταναλώνουν οι φώκες πάρα πολύ σημαντικά είδη αλλιευμάτων, ίσως περισσότερα από αυτά τα οποία εκφορτώνονται και φτάνουν σε εμά τελικά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο από κοινού όλοι να αντιδράσουμε, αλλά αυτό προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της κατάστασης. Οποιαδήποτε λοιπόν πληροφορία έχουμε θα πρέπει να την αξιολογήσουμε και να μην ε, περιοριζόμαστε σε κάποια σχόλια και να θεωρήσουμε ότι ό,τι συμφέρει, ότι μπλέγουν κάποια πράγματα οι γιατί το συμφέρει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις πληροφορίες. Σήμερα νομίζω ότι μας δόθηκαν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε και προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους έλαβαν το λόγο. Ο κύριος Άγκεν θέλει να επανέλθει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις... Ας κάνω μία από τις 20 ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου. Έχω κάποιους αριθμούς όσον αφορά τον ε, αριθμό των ψαριών που καταναλώνουν οι φώκες. Λέει περίπου ότι στη Βαλτική για τον Ο Σολωμός που αλλιεύθηκε και εκφορτώθηκε στην ε, Βαλτική ήταν 340.000 κιλά, όχι τόνοι. Έχουμε 25.000 φώκες και αν τρώει κάθε καθεμία μισό κιλό σολομό την ημέρα θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια σολομού που πρέπει να καταναλώνουν όλες αυτές ε, ετησίως. Τι νούμερα είναι αυτά. Έχω την εντύπωση ότι είναι σωστά, αλλά θα ήθελα να μου τα σχολιάσει κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή. Διότι έχω την εντύπωση ότι οι φώκες καταναλώνουν πολύ περισσότερο το του ε, Σολομού από αυτές οι οποίες φτάνουν ε, στην, ε, και εκφορτώνονται για την ε, δική μας κατανάλωση. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης πέρα και γιατί για μας υπάρχει πρόβλημα στην ακτή ε, Ολλανδία Γερμανία και πιο πέρα. Ε, έχουμε υπολογίσει το μετρήσει τον πληθυσμό η διατροφή είναι 5 ε, κιλά όπως ε, είπατε τη μέρα, όπως ελέγχθη τη μέρα. Εκείνο όμως το οποίο μας δημιουργεί μας πρόβλημα είναι το εξή. Ότι οι αλληλίε μας, μας λένε χρησιμοποιούν ένα κάποιο μοντέλο για το πληθυσμό και την ανάπτυξη του πληθυσμού. Η, μέχρι τώρα ε, το μοντέλο αυτό λέμε, λέει 10% ανά και αυτό το είδαμε να συμβαίνει τα τελευταία τα προηγούμενα χρόνια αλλά όχι τώρα. Ε, επίσης οι αλλοίς λένε ότι ε, μας λένε ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα ποσοστά αλλιευτικών αποθεμάτων εξαφανίζονται, ε, ε, ε, κλείπουν πράγμα το οποίο δεν μπορούν να το αιτιολογήσουν. Δηλαδή αυτή η μη αιτιολογημένη μείωση για ορισμένα είδη, για το γάδο παραδείγματο χάρη, τέτοιου για γαδό είδη, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το μοντέλο αυτό, θα θέλαν πάρα πολύ να καταλάβουν που προ... από πού προέρχεται. Υποψιάζονται όμως ότι προέρχεται και αυτό από τις φώκες, άρα το μοντέλο δεν είναι 100% αξιόπιστο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Και φέρουμε εδώ πέρα σε μια έκθεση της ISIS, μια περσινή έκθεση. Ίσως ο Φιλ Χάμοντ θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό που θα πω. Στην έκθεση της ISIS λέγεται ότι έχουν αυξηθεί από 32.000 έως 40.000 οι γκρίζες φώκες στη Δυτική Σκοτία τις τελευταίες δεκαετίες, τρώνε κυρίως γάδο και η θνησιμότητα του γάδου εξαιτία της στήρευσης της φώκες θα είναι μάλλον σημαντική και αυτό ενδεχομένως να μην επιτρέψει στο απόθεμα γάδου να ανασυσταθεί. Νομίζω ότι η τελευταία αυτή φράση της έκθεσης της ISIS είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να σχολιάσετε το πόρισμα αυτό. Επίσης να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Βέστερμπεργκ. Αν αφαιρέσετε τον σημαντικότερο θηρευτή, ενδεχομένως, προκειμένου τη φώκια, ενδεχομένως να προκαλέσετε την εμφάνιση ενός ενδιάμεσου θηρευτή. και αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε καν τα λεφτικά αποθέματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας με, τον, με τη σειρά που πήραν το λόγο σήμερα το πρωί και να δώσω πρώτα το λόγο στον Φιλ Χάμοντ ζητώντας του να απαντήσει τις ερωτήσεις που έχουν σχέση με τη δική του παρουσίαση, με το δικό τον τομέα. Φιλ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στη δική σας την ερώτηση. Η έκθεση και το πόρισμα της άεσης είναι σωστό. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση του may, ε, ίσως. Για την επίπτωση δηλαδή μπορεί να έχουν ε, οι φώκες την δυνατότητα ανασύστασης ε, του αποθέματος γάδου. Όντως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές γκρίζες φώκες οι οποίες τρώνε μεγάλο ποσοστό γάδου. Ένα μικρό ποσοστό του γάδου έχει μειωθεί εξαιτία τη Έχει μειωθεί λοιπόν κυρίω το απόθεμα, κυρίω λόγω τη φώκια. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα σε μια σύγκρουση τοπική. Οι συνάδελφοι από την Βαλτική μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό περισσότερο. Μιλάω, μιλάω για το γενικότερο πλαίσιο. Όντω, λοιπόν, συμφωνώ με την έκθεση και το πόρισμα τη ISIS, Έτσι έχει η κατάσταση για τις ε, φώκες οι οποίες καταναλώνουν ένα μεγάλο ποσοστό από τον πληθυσμό γάδου. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι τι μπορεί να κάνει κανείς. Και το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που μιλάμε για πληθυσμό φώκες που επηρεάζει έναν ε, μεγάλο πληθυσμό αλίας μεγάλης κλίμακας, η μόνη λύση είναι η θανάτωση μεγάλου αριθμού φωκών. Δεν μπορούμε τοπικά μόνο να θεραπεύσουμε το πρόβλημα σκοτώντας κάποιες φώκες δόθηκήθε πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο πληθυσμός των φωκών προκειμένου να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, μια κάποια αλλαγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η απόφαση είναι σημαντική. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα περιορίσουμε όντω σημαντικά τον αριθμό των φωκών προκειμένου να ανασυσταθεί το απόθεμα γάδου. Πριν από τρει εβδομάδε πήγα σε ένα εργαστήριο στον Ανατολικό Καναδά, όπου ακριβώ το ίδιο ζήτημα συζητούσαν. Λέγανε ότι δεν έχει ανασταθεί ο πληθυσμό γάδου παρουσιάζει μάλιστα ακόμα μείωση σε κάποιε περιοχέ. Αντίστοιχα έχουν αυξηθεί οι φώκε στη ίδια ποσοστά με την Ευρώπη, πάνω κάτω στη ίδια ποσοστά με την Σκοτία. Επομένω, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δουν τι μπορούν να κάνουν και προσπαθούν να πιέσουν οι επιστήμονε στην κυβέρνηση του Καναδά να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του πληθυσμού τη φώκια. Καταλαβαίνετε ότι οι απόψει δίστανται στον Καναδά, ακούστηκαν διάφορε απόψει. Πρώτον, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε ακριβώ πώ θα εξελιχθεί το περιβάλλον αν μειώσουμε τον πληθυσμό τη φώκια και αν θα εμφανιστούν κάποιοι ενδιάμεσοι θηρευτέ, κάποια άλλα αρπακτικά δηλαδή. Πρώτον αυτό. Δεύτερο. ίδια η άποψη τη κοινή γνώμη, τη κοινωνία. Νομίζω ότι η δική σας η Επιτροπή θα πρέπει να το εξετάσει και να το συζητήσει αυτό. Πρέπει πραγματικά να μειώσουμε δεκάδες χιλιάδες, να σκοτώσουμε δεκάδες χιλιάδες φώκες, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός, πληθυσμός τους και να σταθεί το λευτικό απόθεμα. Η άποψή μου είναι ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, κινδυνεύουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ούτε καν αν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμφωνώ λοιπόν με το πόρισμα της ISIS, αλλά εκκρεμεί ακόμα το ερώτημα του τι μπορούμε να κάνουμε και το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό. Οι συνάδελφοι από τη Βαλτική θα μπορούσαν να πούνε περισσότερα πράγματα. Πάντως στην Σκοτία Ανεπίσημα αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι αν υπάρχουν φώκες που επηρεάζουν σε τοπικά εντοπισμένες ζώνες την υδατοκαλλιέργεια ή την μικρού κλίμακας αλίας σε συγκεκριμένες παράκτης ε, περιοχές, τότε ναι, υπάρχει άδεια για το κυνήγι και την θύρευση της φώκιας. Σε τοπικό λοιπόν επίπεδο κάτι μπορεί να γίνει, αλλά σε γενικότερο επίπεδο δεν νομίζω ότι μπορεί πραγματικά μέσω του πυροβολισμού της φώκιας να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Όπως σας είπα, έχουμε ένα νέο νομοθέτημα στη Σκοτία για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, όπου αναγνωρίζεται το πρόβλημα αυτό του πληθυσμού της φώκιας, αλλά λέγεται ότι θα πρέπει να διευθετηθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η Σκοτία κινείται σωστή κατεύθυνση και ότι ναι, μεν σε τοπικό επίπεδο το πρόβλημα λύνεται με τον πυροβολισμό, σε ένα ευρύτερο επίπεδο ο πυροβολισμός, η θανάτωση αυτή της φώκιας δεν μπορεί να έχει αναγκαστικά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο κύριος Άγγλαντ από τη Φινλανδία μίλησε για την κατάσταση στη Βαλτική και ανέφερε ορισμένες επιδράσεις ε, που υπάρχουν, συνέπειες που υπάρχουν που δεν είναι σωστές κατά την άποψή μου. Δεν ε, Νομίζω ότι ο πληθωσμός της Φώκιας αυξήθηκε υπέρμετρα στη Βαλτική τα τελευταία χρόνια. Το 2000, μέχρι το 2006 ε, κάποιο είδος Φώκιας αυξανόταν και μετά σταθεροποιήθηκε. Τώρα για τις ριγέ φα, ε, ε, τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά από το 88 και δόθε η αύξηση του πληθυσμού της, ε, ε της ριγέ αυτής φώκιας ε, αν θέλετε είναι στο 50% του ρυθμού ανάπτυξης των άλλων πληθυσμών 180.000 άτομα ριγέ Φώκε υπάρχουν ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στη δεκαετία του 20 και του 30 ε, σκοτώνονταν ε, κάθε χρόνο 10 με 15 φω, τέτοιες φώκες. Αλλά Ε, και τώρα βεβαίως ε, θανατώνονται φώκες 2-3 ε, χιλιάδες το χρόνο αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική εν πάση περιπτώσει για, και για την κρίζα φώκια ε, υπήρχε μια αύξηση τα παλιά τα χρόνια αν θέλετε που πρόσφατα δεν συνεχίζεται και για τις βαλτικές χώρες ε, δεν υπάρχει αυτή η υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού που ανέφερε ο Φινλανδός ο συνάδελφός μας εδώ ε, στην ICS υπάρχουν στοιχεία και μπορείτε να τα βρείτε. Βεβαίως, ε, μέχρι το 2006 υπήρχε μια αύξηση κατά 8,5 περίπου τα 100 γενικώ του πληθυσμού της Φώκιας, αλλά όχι μετά το 2006. Εκεί υπάρχει σταθεροποίηση. Τώρα για τις ποσότητες τροφής που καταναλώνουν ή τα διάφορα είδη φώκιας δεν έχουμε πολλά στοιχεία, αλλά έχουμε στοιχεία για συγκεκριμένες τοποθεσίες, συγκεκριμένες περιοχές που όμως δεν μπορούμε μετά να τις ε, να επεκτείνουμε και να τις γενικεύσουμε και να πούμε ότι αφορούν σε ολόκληρο το πληθυσμό της γκρίζας της φώκιας. Η... Έχουμε τρία είδη φώκιας όπως είπαμε και τα τρία αυτά είδη φώκιας έχουν διαφορετικές συνήθειες. Είπαμε, οι ριγέ φώκε δεν αυξάνονται στον κόλπο της Ρίγκα ή στην Φινλανδία. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τα πράγματα. Πόσα ψάρια τρώνε φώκες στη Βαλτική. Δεν είναι εύκολο το ερώτημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν ξέρω εδώ, ο συνάδελφος μπορεί να μας δώσει περαιτέρω στοιχεία. Αλλά και μάλλον ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που ελέγχθησαν. Απειλές κατά του των της Φώκιας. Στη Βαλτική, για τη Ριγέτη Φώκια, αυτή ζει στη Βαλτική μόνο και μόνο επειδή υπάρχει πάγος. Αλλά οι πάγοι τα τελευταία 20 χρόνια φθήνουν, όπως ξέρετε. Και στο νότο, ας πούμε, στο κόλπο της Ρήγας η ρυθμή ανάπτυξη του πληθυσμού της Ριγέ Φώκιας ήταν αρνητική. Η άλλη είναι η κατάσταση για την κρίση φώκιας, γιατί έχουν γίνει περισσότερες μελέτες εκεί. Κάναμε μελέτες για τη θνησιμότητα ε, και για τη θνησιμότητα των νεογνών στη Βαλτική και είδαμε ότι η θνησιμότητα για τους, τα νεογνά τον πρώτο χρόνο έφτανε τα 30% όταν αναγκάζονταν να γεννήσουν όχι σε πάγο αλλά σε ε, στη γη, σε χέρσο. Ε, μεγάλη φθηνισμότητα λοιπόν κατά την πρώτη διάρκεια ζωής. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι μειώνεται ο πάγος στη Βαλτική Οπότε τα νεογνά πεθαίνουν περισσότερο γιατί γεννιούνται, είναι αναγκασμένες οι μητέρες να γεννήσουν σε, στη γη, στη χέρσο. Επίσης υπάρχουν μολύνσεις οι οποίες επηρεάζουν την θνησιμότητα των νεογνών. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν με την μείωση των, των πάγων επηρεάζει και τον πληθυσμό της Φώκιας. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν μη αιτιολογημένες μη απώλειες αλλά συνέβησαν και πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Το 1990-91 πέθανε το 50% του πληθυσμού της Ριγέ Φώκιας στον κόλπο της Ρήγας. Δεν ξέρουμε γιατί αλλά μοιραία βγάζουμε μέσω όρου, μέσους όρους και οι μέση όροι αναφέρονται στην περίπτωση που δεν ε, συνέβη ένα καταστροφικό γεγονός. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ε, καταστροφικά γεγονότα. Η πιθανότητα της ύπαρξης ε, καταστροφικών γεγονότων μπορεί να είναι πολύ ψηλή, αλλά δεν τα υπολογίζουμε αυτά τα καταστροφικά γεγονότα όταν βγάζουμε μέσους όρους. Μέσους όρους βγάζουμε αφαιρουμένων των καταστροφικών γεγονότων. Επίσης, για τις φώκες στη Βαλτική. Η κατάσταση αλλάζει και για την κρίζα φώκια και για τη ριγέ φώκια η κατάσταση υγείας των ζώων ε, επιδεινώνεται όπως ελέγχθη το πάχος του λίπους ε, της στιβάδας ε, του λίπους μειώνεται και αυτό δεν είναι καλό επίσης α, αυξάνονται τα α, έλκη του ε, ε, στο, κολονικά ε, έλκη το οποίο οφείλονται σε συγκεκριμένα ε, σκουλίκια. Σκουλίκια τα οποία μπορεί να είναι αποδολώματα αγκιστριών χρησιμοποιούνται μέχρι οτιδήποτε άλλο. Ε, επίσης η αναπορική παραγωγική υγεία των ζώων αυτών επιδεινώνεται. Υπήρξαν αλλαγές στα, τα, τελευταία χρόνια παραδείγματο χάρη στο κατεγάκι, κατεγάτι είχαμε 12% αύξηση μέχρι πριν από μερικά χρόνια και τώρα πέσαμε στο 3% αύξηση. Άρα τα παλιά σενάρια και μοντέλα με εκθετικού όπου η αύξηση θα ήταν εκθετική διαχρονικά ε, αυτά δεν ισχύουν πια. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πια σωστές διότι οι υποθέσεις εργασίας ήταν λάθος. Τώρα για, για την κοινή φώκια μετρήθηκαν στις περιοχές που αναφέρθηκαν 22.000 άτομα το 88, το 2002 όμως υπήρχαν, ε, συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία, τα επηρέασαν ε, τον πληθυσμό. Τα τελευταία χρόνια όμως ε, δεν υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, μεγάλες καταστροφές. Σταθεροποιήθηκαν τα πράγματα και για το μέλλον δεν μπορούμε να αναμένουμε τουλάχιστον στο βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό ε, αύξηση του πληθυσμού της φώκιας. στις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αλή, παράκτη αλία μικρής κλίμακος που να χρησιμοποιεί τι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Βαλτική. στη Βαλτική αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται όταν δεν υπήρχαν πολλές φώκες παραδοσιακές μέθοδοι ας πούμε και τα λοιπά. Τώρα ίσως επειδή αυξήθηκε αλλά όχι υπέρμετρα ο πληθυσμό της φώκιας τώρα γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν ναι, ε, ευξημένα προβλήματα. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ λέει ε, ο πρόεδρος η κυρία Κρόνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ για να απαντήσει τον κύριο Χάγκλιν για τον έλεγχο τον πληθυσμό. Εμείς δεν έχουμε, όπως σας είπα, ε, πάρα πολλά αποδεκτικά στοιχεία για τους πληθυσμούς που υπάρχουν στα δικά μας τα είδατε, τα Ιρλανδικά και τον συσχετισμό. Έχουμε πάρα πολύ λίγες πληροφορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν συμβαίνουν, αλλά βλέποντας ε, τις, ε, το μέγεθος του πληθυσμού σε στέλνουμε άλλες παράκτιες περιοχές, πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε λίγες. Και σε σχέση με το τι έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς έχουμε για την ε, φώκια την κοινή 5% φερρυπίν, 6.000 περίπου. Και κάτι ανάλογο για την γκρι. Βεβαίως, τα στοιχεία που έχουμε είναι από, τις, από τους αλληλείς που χρησιμοποιούν τα σταθερά εργαλεία. Και εκεί μιλούμε για απώλειες 10%. Τώρα όσον αφορά την ε, πελαγική αλία και τις ε, μεγάλες τράτες τις οποίες χρησιμοποιούν ολίγοι για να αλλιεύουν οι μεγάλες οι οικογένειες δεν έχουμε στοιχεία και εξάλλου θα ήταν ίσως περιθωριακά. Δεν ξέρουμε σχετικά με το σύνολο των αλλιευωμένων ειδών απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό της. Και θα πρέπει να κάνουμε, όπως είπα και προηγουμένως, μελέτες και σαφείς εκτιμήσεις όλοι από κοινού για να βρούμε μία λύση. Προστημονική, ακαδημαϊκή κοινότητα, εκπαινήσεις και τα λοιπά. Τώρα, σε σχέση με την ε, κατάσταση και την κατάσταση υγείας των θηλαστικών, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, ούτε για τις τάσεις που επικρατούν, Άρα δεν γνωρίζουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε από τα διάφορα στοιχεία που υπάρχουν ότι υπάρχει κάποια αύξηση σε κάποιες περιοχές. Σε εθνικό επίπεδο όμως δεν έχουμε στοιχεία. Έχει φύγει ο κύριος Γκάλαχερ, είπε όμως προηγουμένως ότι η τελευταία απογραφή έγινε το 2003-2005 και από τότε δεν έχουν γίνει τίποτε πιο τελευταία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να κάνουμε κάποια εθνική απογραφή ε, του χρόνου σε δύο χρόνια για να δούμε αν υπάρχει κάποια ε, αλλαγή, κάποια αύξηση σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία έχουμε το 2003. Έχουμε κάποια μικρά στοιχεία όσον αφορά τα παράσιτα, τα διάφορα ε, σκουλίκια τα οποία προσβάλλουν την υγεία της φώκιας. Οι Ιη που τους προσέβαλαν τον δεκαετία του 80 και του 90 ε, δεν επηρέασαν πάρα πολύ το συνορικό πληθυσμό και από όσο καταλαβαίνουμε η μεγαλύτερη ε, καταστροφή προκαλείται κυρίως από τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα και από διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με μελέτη που έγινε τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια εθνικής εμβέλειας μελέτη. Και βεβαίως η παράνομη, ε, παράνομο κυνήγι από τους αλείς είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια κοινή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και όπως σας είπα προηγουμένως με μια πιλωτική με λέτη στην Δυτική Ιρλανδία και με το ότι θα έχουμε κάποια άτομα που θα εποπτεύουν τα όλα συστήματα επάνω στα αλλιευτικά σκάφη θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα και τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι πρακτικές για να μπορέσουμε ακόμη και να βελτιστοποιήσουμε τις αλλιευτικές πρακτικές. Αυτό είναι ε, κάτι με το οποίο έχουν συμφωνήσει και οι αλληλείς ε, και για, θα μας επιτρέψει να έχουμε στοιχεία που θα αφορούν και την παρεμπίπτουσα αλληλεία και να ξέρουμε και τον αριθμό τον ακριβή των θηλαστικών που φτάνουν και στις ακτές. Ευχαριστώ. Τελικά ο κύριος Βέστεμπεργκ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής για την κατάσταση στη Βαλτική. Εγώ προσπάθησα να κάνω κάποια γενικά ε, σχόλια όσον αφορά το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ φώκιας και αλίας. Για την ε, Βαλτική θα πρέπει να έχουμε κατά νου ποιες είναι οι ζημίες που προκαλούνται για τους αλίες, για την αλία γενικότερα. Και να έχουμε και ε, κατά νου ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες ε, ε ζημίες που προκαλούνται κυρίως την παράκτη αλία στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, πολλοί αλληλείς δεν μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους διότι προκαλούν τρομερές ζημιές ή φώκες. Ζημιές στα δίχτυα, στα αλλιεύματα, πράγμα το οποίο εξηγεί ότι και το κυνήγι της φώκιας έχει επιτραπεί για να μπορέσουν να αντισταθμιστούν οι ζημιές που προκαλεί. Βεβαίως δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη μαρτυρία ή απόδειξη όσον αφορά τις ε, βλαβερές επιπτώσεις αυτού του κυνηγιού κατά της φώκιας erfarenheten av skyddsjakt på knubbsäl är att det kan ha betydande effekt. Både då när det gäller eh, skador på... på... Έχουν κάποια είδη φώκες που είναι αυτά τα οποία προκαλούν τις περισσότερες ζημιές κυρίως στην παράκτη αλία και που προκαλούν ζημιές και στις διάφορες ε, εγκαταστάσεις της ε, υδατοκαλλιέργειας. Φαίνεται ότι οι γκρίζες φώκες είναι λιγότερο επιθετικές. Άκουσα την κυρία Λέβινγκ, αυτά τα οποία είπε είναι ενδιαφέροντα. Αλλά είναι σαφές ότι εάν μετακινηθούν οι, οι φώκες, επανέρχονται ούτως ή άλλως. Και βεβαίως, εάν τις μετακινήσουμε, θα έχουμε να κάνουμε με άλλα αρπακτικά, με άλλους τυρευτές, οι οποίοι ποιοι θα είναι και τι κακό θα προκαλέσουν. Όσον αφορά τα αλλιευτικούς πόρους έχω κάποια διαφορετική εκτίμηση από τη δική σας. Έχουμε όμως πολύ λίγα στοιχεία στη διάθεσή μας. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι επιβλαβείς επιπτώσεις της ε, ε, φώκιας για το Σολομό Φερρυπίν είναι πολύ περισσότερες από ό,τι για άλλα αλλιεύματα. Έχουμε όμως, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ λίγα στοιχεία. Υπάρχουν πολλά κενά, δεν έχουμε ακριβή δεδομένα και έτσι δεν έχουν τελικά καμία πραγματική αξία όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ε, γίνει μέτρηση βάσει των ε, κομματιών των ψαριών που βρίσκουμε. Βρίσκουμε κόκαλα, βρίσκουμε το κεφάλι του ψαριού, αλλά πολλέ φορέ δεν ξέρουμε ποιο κόκαλο αντιστοιχεί σε ποιο κεφάλι. Αλλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε εύκολα τα είδη τα οποία προτιμούν οι φώκες. Και το κυνήγι που επιτρέπεται στην Βαλτική δεν επηρεάζει την κατάσταση τελικά. θα έπρεπε να θανατώνονται τουλάχιστον 2 με 3 χιλιάδες άτομα ετησίως για να ξέρουμε τι γίνεται. Πράγμα το οποίο όμως δεν μπορεί να συμβεί. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι όταν συγκρίνεται ένα συγκεκριμένος αριθμός στηλαστικών βάσει των στοιχείων ε, που έχουν αυτοί που τα κυνηγούν, δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα. Έχουμε ένα ενσταντανέ, αν θέλετε, κάποια στιγμή μία εικόνα, μία συγκεκριμένη στοιχή. Στιγμή. Αλλά δεν έχουμε πιο έγκυρα στοιχεία. Και αν συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία με τον αριθμό των ε, ζώων που έχουν μετρηθεί, θα μπορούσα να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προβολή, διότι δεν είναι συγκεκριμένα και τα στοιχεία που έχουν. Ε, Ένα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 Ε, ακούσαμε να αναφέρονται παραδοσιακές μέθοδοι αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι ήταν εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν είχαμε 300.000 φώκες πληθυσμό άρα δεν μπορεί να είναι σωστή αυτή η προσέγγιση και ένα άλλο ερώτημα το οποίο ετέχει ετέθη με συγχωρείτε ε, σχετιζόταν με άλλα αρπακτικά άλλους θηρευτές. Δείτε, ο κύριος θηρευτής είναι η φώκια. Υφίσταται, αυτό είναι γεγονός. και άπαξ και και υπάρχουν πολλοί άνω του ενός θηρευτές εκ των οποίων ένας είναι κύριος οι υπόλοιποι θηρευτές κυνηγούν τον κύριο θηρευτή καθώς καταλαβαίνετε γι' αυτό άμα αφαιρέσει κανείς τις φώκες ως κύριο θηρευτή το, ο δευτερεύον θηρευτής παραδείγματος χάρη ε, παίρνει τη θέση του κυρίου θηρευτή. Αυτό προσπαθούσα να πω όταν έλεγα ότι δεν αλλάζει κατάσταση αν αφαιρέσουμε τις φώκες δεν εννοούσα ότι οι φώκες δεν είναι θηρευτές και δεν έχουν επιδράσεις απλώς το ψάρι ή το θαλασσοπούλι που είναι ο υπαριθμόν δύο θηρευτής αντικαθιστά τη φώκια που είναι ο υπαριθμόν ένα Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι προς το παρόν για τα, για τα αλλιευτικά αποθέματα ο κύριος θηρευτής αν μπορώ να το ονομάσω έτσι ή το κύριο ε, κυρίως ένοχη είναι η αλία. Ε, ε, από αυτούς, από τους κι μας κινδυνεύουν τα λευτικά αποθέματα. Εκεί όμως μπορούμε να ε, διαχειριστούμε τα πράγματα και να επέμβουμε. Α, δεν μπορούμε να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο για τη φώκια ως ε, ένοχο για τη μείωση των αλληλευτικών αποτελεσμάτων και σίγουρα δεν είμαστε τόσο ε, σίγουροι για τα στοιχεία ούτως ώστε να μπορούμε να διχειριστούμε καλά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Βέστερμπερκ. Ο κύριος Χάμον θέλει να πάρει το λόγο, θα μιλήσει και αυτός ειδικά. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ε, έχετε δίκιο. Η πρόκληση είναι πολύ σημαντική. Το πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τις φώκες. Το θέμα δεν είναι να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τον υψηλότερο δυνατό αριθμό των φωκών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να δούμε πώς απειλείται από τις φώκες η δική μας επαγγελματική αλία. Έχουμε την έκθεση του ISIS που μας λέει ότι θα έχουμε αύξηση της τάξης του 20-30% ε, τα επόμενα χρόνια. τα δικά μου δεδομένα βέβαια, μάλλον αν κοιτάξουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι τα δεδομένα θα κινηθούν κάπως διαφορετικά. Όσον αφορά δηλαδή πάντα τις επιπτώσεις ε, των φωκών στην Αλία. Είχαμε μια αύξηση 15% πέρυσι για την κρίζα φώκια στην ε, Φιλανδία. Για την κοινή φώκια ή την φώκια με τις ραβδόσεις δεν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα στη χώρα μου. Έχουμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα, όπως βλέπετε, για τις γκρίζες φώκες, που ακόμα και αυτές όμως επιφέρουν πολλά προβλήματα στην επαγγελματική αλληλεία. Η πρόθεσή μας λοιπόν δεν είναι να διαχειριστούμε προς το δικό μας συμφέρον το οικοσύστημα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά η οπτική γωνία, η σκοπιά αλλάζει με βάση το που στεκόμαστε κάθε φορά πώς προσεγγίζουμε δηλαδή το ζήτημα. Το σεμινάριο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα και με ηλεκτρονική μορφή για να καταφέρουμε να εξετάσουμε όλα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα και για να καταφέρουμε να εξολογήσουμε περισσότερο όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν για τον πληθυσμό. Θα ήθελα λοιπόν πολύ ή δυνατόν μετά το τέλος της συζήτησης να μας στείλετε ηλεκτρονικά όλες αυτές τις παρουσιάσεις, όλες αυτές τις πληροφορίες, ιδίως αυτές που έχουν να κάνουν με αριθμητικές παραστάσεις και δεδομένα. Σας ευχαριστούμε. But, okay, distribute, uh, Ναι, ναι, προφανώς θα σας δώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και επιπλέον πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ακρόαση αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μιλητές για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν. Η λύση θα ήταν ε, να χρησιμοποιήσουμε τηλεμετρικές μεθόδους για να καταφέρουμε να εντοπίσουμε, αν θέλετε, όλες αυτές τις ε, φώκες, λέει αστευόμενος ο Πρόεδρος. Ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να έλυνε το πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χάρκονεν, τον κύριο Χάμοντ, την κυρία Κρόνιν και τον κύριο Βέστερμπερκ για την πολύτιμη συμβολή τους και για τις απαντήσεις που δώσανε στα μέλη της Επιτροπής Ελίας. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Ας περάσουμε τώρα στα διάφορα. Επιθυμεί να πάρει κανείς το λόγο στο σημείο αυτό. Δεν έχουμε κανένα σημείο, επομένω περνάμε στο σημείο 10, ανακοινώσει τη Προέδρου σχετικά με τι αποφάσει που λαμβάνουν οι συντονιστέ. Νομίζω ότι ήταν μία από τι πιο εύκολε συνεδριάσει συντονιστών που είχαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εδώ συγκεκριμένε αποφάσει για να ανακοινώσουμε. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει στι Βρυξέλλε στι 30 Νοεμβρίου, 3 το μεσημέρι έω 6.30 και την 1η Δεκεμβρίου 9 το πρωί έω 12.30 και 3 έω 6.30. Για όσους περιμένουν βέβαια ακόμα και μπορούν να παραμείνουν, θα προβάλλουμε το έργο της WWF, το οποίο συζητήσαμε εκτενώς χθες στη συνεδρία της Επιτροπής. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι της WWF είναι εδώ και μπορούν να αρχίσουν με την προβολή της ταινία. Μου ζήτησαν επίσης να πω κάποια λόγια εν είδη εισαγωγής. Καταρχάς λοιπόν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας ε, εδώ, για το ότι ήρθατε να δείτε το ντοκιμαντέρ αυτό. Προβλήθηκε το Σαββατοκύριακο το αυτό, ενδεχομένως να το είδατε κάποιες στις χώρες σας. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι το πόρισμα μιας έρευνας που διέρχησε 7 ε, μήνες της ICIJ με ένα κανάλι το οποίο δικαίβεται σε ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον προβλήθηκε στο πρόγραμμα του BBC Life on the Edge και αποτέλεσε βάση κάποιων άρθρων που είδαμε στους Sunday Times, στην Le Soir και στον ε, EU Observer. Ότι φαίνεται θέλουν να ξεκινήσουν ε. και θα εμφανιστούν και πολλά άλλα άρθρα και σε άλλες ε, ευρωπαϊκές εφημερίδες. 11 δημοσιογράφοι λοιπόν κάνανε 200 περίπου συνεντεύξεις με αλληλείς, ε, διάφορους αξιωματούχους, επιστήμονες και ανέλησαν ε, πάρα πολλά έγγραφα δικαστηρίων καθώς επίσης και πάρα πολλές εκθέσεις και κανονισμούς. Και στο ντοκιμαντέρ αυτό μας λένε ότι έχουν ανακαλύψει ένα πολύ μεγάλο επίπεδο ε, παρατυπιών κακής διαχείρισης που αντιστοιχεί σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια ένας στους τρεις ερυθρούς ε, τόνους δεν καταγράφεται στο μερολόγιο του πλοίου μεταξύ 1998 και 2007 και το εικονικό αυτό είδος, λένε, το συμβολικό αυτό είδος βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, της εξαφάνισης. Την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι θα γίνει συνεδρίαση της ΆΙΚΑΤ, επομένω θεωρώ ότι το ντοκιμαντέρ αυτό προβάλλεται την κατάλληλη στιγμή για όσους ήταν ε, εδώ και χθε. Ξέρετε ότι ακούσαμε τον κύριο Κώστερ, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλίας του Βίγκο, ο οποίος μας έκανε μια πολύ λεπτομεριακή παρουσίαση της κατάστασης για τον ερυθρό τόνο. Μας είπε ότι επικεντρώθηκαν στο είδος αυτό τα τελευταία τρία χρόνια και σε απάντηση πολλών, σε πολλούς συναδέλφους οι οποίοι αναφέρθηκαν στα άρθρα αυτά και στο ντοκιμαντέρ αυτό, ο κύριος Κώστερ είπε ότι οι πληροφορίες του ντοκιμαντέρ είναι ακριβείς για την περίοδο 2006-2007. Αλλά είπε ότι ε, οι δραστηριότητες υπηρεσίες επιτήρησης έκτοτε έχουν ε, βελτιωθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους 12 μήνες. Συνεπώ ελπίζω ότι οι βελτιώσεις αυτές θα συνεχιστούν και ελπίζω ότι τα όσα θα δούμε τώρα στο ντοκιμαντέρ δεν ισχύουν πλέον. Πάντως το ντοκιμαντέρ αυτό μπορεί να συμβάλλει στην όλη συζήτηση που έγινε και θα πρέπει να το δούμε εν ώψη της συνεδρίασης της ICAT στο Παρίσι. Ας προσπαθήσουμε και μια τρίτη φορά τώρα να ξεκινήσουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ. But what changes our lives changes nature too. Globalizing how we use nature's resources needs global cooperation. But as this story shows, that can be a long time coming, if it comes at all.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 Ευχαριστώ πολύ και το WWF για το που μας ε, έκανε αυτή την προβολή